Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, επιτρέψτε μου καταρχάς να σας ευχαριστήσω που δεχτήκατε να συμμετάσχετε στην συνάντηση αυτή που αφορά στις σχέσεις ανάμεσα στις γυναίκες και την Ευρωπαϊκή Ένωση εν ώψη των ευρωεκλογών του 2014. Η σημερινή μας συνάντηση αποτελεί το σημείο εκκίνησης των δραστηριοτήτων που πρόκειται να αναπτυχθούν και αναλυθούν από το Ευρωκοινοβούλιο σχετικά με την Διεθνή ημέρα της γυναίκας στις 8 η Μαρτίου. Λοιπόν, στόχος ε, για την έναρξη αυτών των σειράς των εκδηλώσεων είναι διτός. Να τονίσουμε την συμβολική σημασία αυτής της διεθνής, διεθνούς ε, παράλληλα προσφέροντας ε, μία σειρά από ενημερώσεις για θέματα που αφορούν τις σχέσεις ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις γυναίκες. Επιτρέψτε μου να αναφέρω σε μερικές αυτές τις εκδηλώσεις. Πρώτα απ' όλα η ομιλία που θα γίνει από τον πρόεδρο μας Γιώργη Μπούζεκ την 8η Μαρτίου άμα την άρξη της συνόδου στο Στρασβούργο. Ε, εν συνεχεία θα υπάρξουν διάφορες εκδηλώσεις που θα αφορούν την καταπολέμηση της βίας που ασκείται ενάντια στις γυναίκες και ιδιαίτερα η συνεδρίαση που θα διεξαχθεί την 16η Μαρτίου στο ημικύκλιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εδώ στις Βρυξέλλες με την συμμετοχή των ομολόγων μας από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Κυρίες και κύριοι, τις τελευταίες ημέρες οι διάφορες έρευνες που έχουν γίνει περί του θέματος αποκαλύπτουν πως η σχέση ανάμεσα στις γυναίκες και την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι λιγότερο ισχυρή από αυτήν που συνδέει την ε, άνδρες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά διάρκεια λοιπόν αυτής της ημερίδας θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε το ζήτημα. Ποια είναι η φύση αυτών των σχέσεων, ποιες ε, και τι μπορούμε να κάνουμε και πώς μπορούμε να ενισχύσουμε αυτή τη σχέση Ίσως ε, θα πρέπει να αναρωτηθούμε εάν στις διάφορες έρευνες οι άνδρες και οι γυναίκες ε, απαντούν με την αυτή ειλικρίνεια στα ερωτήματα που τους τίθενται. Αλλά αυτό δεν είναι ο στόχος της σημερινής μας συναντήσεως. Πάντως ε, τα ερωτήματα αυτά, τα αποτελέσματα αυτά μας αφορούν άμεσα. Γι' αυτό λοιπόν είναι επιτακτικό να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια προκειμένου να προσεγγίσουν οι γυναίκες περισσότερο την Ευρωπαϊκή Ένωση καταδεικνύοντάς τους ποιε είναι οι επιπτώσει στην καθημερινότητά τους και πως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι φορέας ενός προγράμματος, ενός οράματος ε, τόσο για τις γυναίκες όσο για τους άντρες. Μπορούμε έτσι να ενισχύσουμε την κινητοποίηση του εκλογικού σώματος των γυναικών κατά τις εκλογές του 2014. Για να το πετύχουμε χρειάζεται να πάμε ακόμα παραπέρα από ότι διάφορες εκδηλώσεις, οι ορθασμοί, οι μερίδες που υπερθυμίζουν την ισότητα των φίλων. Να μην παρεξηγηθούν τα λόγια μου, πάντως η κινητικότητα γύρω από την ημέρα της γυναίκας ε, την 8 Μαρτίου είναι κάτι το απαραίτητο και ε, με ιδιαίτερο συμβολισμό, αλλά δεν επαρκεί. Αυτή η συνάντηση για μας θα πρέπει να αποτελέσει την ευκαιρία για να κάνουμε την διάγνωση, να αναλύσουμε τις αιτίε και να ασχοληθούμε με τις δράσεις που πρέπει να αναλάβουμε έτσι ώστε η ισότητα των φύλων να πραγματοποιείται μέρα με τη μέρα και να δώσουμε μεγαλύτερη προβολή στις δράσεις μας χρειάζεται επιτακτικότατα να βασίσουμε την πολιτική επικοινωνία σε μακροπρόθεσμα προγράμματα καταδεικνύοντας την ισότητα των φύλων και όχι μόνο είναι παρούσα στο πνεύμα μας και στα κείμενά μας αλλά και στις συγκεκριμένες δράσεις μας. Προτού να προχωρήσουμε στη συζήτηση θα ήθελα να τονίσω κάποιες πτυχές που θεωρώ θεμελιώδες πρώτα απ' όλα σε σχέση με την συμμετοχή των γυναικών στις τελευταίες ευρωεκλογές. Θέλω να σχετικοποιήσω την ε, δήλωση σύμφωνα με την οποία οι γυναίκες ε, έχουν, είχαν λιγότερη συμμετοχή από ότι οι άνδρες. Αυτή η εντύπωση πολύ συχνά δίνεται τόσο μέσω των μέσων ενημέρωσης όσο και από ορισμένους αναλυτές. Με όλα τα αυτά οι γυναίκες ψήφισαν στο ίδιο ποσοστό με τους άντρες, δηλαδή 42% έναντι 44%, δηλαδή μια διαφορά της τάξης ε, των δύο μονάδων. και σε οκτώ χώρες θα έλεγα ότι οι γυναίκες ε, ε, πήγαν στις κάλπες ε, κατά μεγαλύτερο ποσοστό από τους άντρες. Αυτό συνέβη και στις εθνικές εκλογές όπου μέσω σε όρος συμμετοχής ήταν ακριβώς ο ίδιος τόσο για τις γυναίκες και για τους άντρες και έφτασε το 72%. Μπορούμε να αναρωτηθούμε λοιπόν εάν αυτός ο τρόπος για την αναφορά στο γυναικείο εκλογικό σώμα δεν αποτελεί μια διακριτική μεταχείριση ε, συνειδητή θα έλεγα και ηθελημένη. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό η κυρία Μπανσουσί θα το καταδείξει και δεν ε, θα πρέπει να εκπλησόμεθα ε, το ότι τα μέσα ενημέρωση δεν αντιμετώπισαν γυναίκες και άνδρες εκλογής με τον αυτό τρόπο. Ε, παρά όλα αυτά τα εμπόδια, γυναίκες αποτελούν σήμερα το 35% των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έναντι 24% στο σύνολο των Εθνικών Κοινοβουλίων. Για να ε, μετρήσουμε τις ε, πρόοδους που έχουν επιτευχθεί αρκεί να θυμηθούμε πως ε, τα ποσοστά αυτά κατά τη διάρκεια των πρώτων εκλογών του 1979 στο Ευρωκοινοβούλιο έφτασαν στο 17 μόλις τα 100 για τις γυναίκες. Βρισκόμαστε λοιπόν πολύ μακριά από την ισότητα. Ενώ οι γυναίκες είναι πιο πολυάριθμες από ότι οι άνδρες στο πλαίσιο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπενθυμίζω πως αποτελούν το 51% έναντι 41% των ανδρών και εμείς ε, ακούμε να λέγεται ότι οι γυναίκες είναι λιγότερο ευρωπαϊστές από ότι οι άνδρες. Σύμφωνα με τα, ποσοστά αυτό το ζήτημα θα πρέπει να το ε, αναλύσουμε. Η παρουσία του κυρίου Στάμφερ θα μας επιτρέψει να το συζητήσουμε. Οι γυναίκες δεν είναι καθόλου μακριά από την Ευρώπη. Είναι ευρωπαϊστές ε, και αναφέρουν ότι δηλώνουν πως ενδιαφέρονται περισσότερο για την ε, πολιτική τόσο τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο από ό,τι σε ευρωπαϊκό. Και αυτό οφείλεται στο ότι πολύ περισσότερο από ό,τι άντρε διαχειρίζονται την ε, οικογενειακή καθημερινότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τους φαίνεται κάπως γραφειοκρατική, τεχνοκρατική και περίπλοκη οι επιπτώσει οι άμεσε ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην καθημερινότητά του και στην καθημερινότητα των οικογενειών του δεν τους έχει εξηγηθεί επαρκώς. Όλοι λοιπόν φέρουμε μια ευθύνη σε αυτό το θέμα και για αυτό το αποτέλεσμα. Οι γυναίκες δεν είναι ότι δεν έχουν το ίδιο όραμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση από ότι οι άνδρες και γι' αυτό είναι λιγότερο ευρωπαϊστρίες. Υπάρχει διαφορά στον τρόπο με τον οποίο αισθάνονται Ευρωπαίες πολίτες. Και γι' αυτό είναι υπέρ της ευρώ και μιας κοινή εξωτερικής πολιτικής, αλλά λιγότερο από ό,τι άντρε. του αντίον όμω επιθυμούν περισσότερο από ό,τι άντρε την ανάπτυξη πολιτικών που αφορούν την εκδήλωση της αλληλεγγύη, όπως η δημόσια υγεία ή και την κοινωνική πολιτική. Υπό το φως λοιπόν της δημοσιονομικής κρίσης και με τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις που αυτή έχει, δεν θα πρέπει να μας εκπλήσει που οι γυναίκες επιθυμούν να προαχθεί αυτή η πολιτική της αλληλεγγύης. Οι ανισότητες σε ζητήματα απασχόλησης και ε, συνολικής ένταξης στην οικονομική ζωή αποτελούν αναφίβολα τις πρώτες αιτίες. Για τον λόγο λοιπόν αυτό επιτρέψτε μου κυρίες και κύριοι να ε, πάρω ένα παράδειγμα. Το ποσοστό ε, απασχόληση των γυναικών είναι χαμηλότερο από ότι των ανδρών. Ανέρχεται σε 59,1% έναντι 72,8% των ανδρών. Δηλαδή έχουμε μια διαφορά της τάξης του 13,7% ποσοστιών μονάδων. Φυσικά η διαφορά είναι πολύ σημαντική, αλλά η διαφορά αυτή μειώνεται σημαντικά έτος με έτος από 2001 όπου η ποστά ήταν 50,4 και 70,9% για τους άνδρες. Δηλαδή η διαφορά ήταν γύρω πάνω από 20%. Θα ετοιμήσετε λοιπόν ότι ο στόχος της της Λισαβόνας για το 2000 ε, για την γυναική απασχόληση ήταν να επιτευχθεί το 60% για το 2010. Περίπου το φτάσαμε, το κουμπάμε αυτό το ποσοστό. Και θα πρέπει να εξηγήσουμε πως ε, χάρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματική πρόοδος έχει επιτευχθεί. Θα χρειαστεί λοιπόν να πείσουμε πως ε, μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα για να καλύψουμε αυτό το χάσμα των διαφορών. Ε, επίσης θα ήθελα να ασχοληθώ με την μισθολογικές διαφορές, μισθολογικό χάσμα που είναι αιτία των ανισοτήτων και της απογοήτευσης. Το 2007 η διαφορά το μισθολογική ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες ε, ανήκει το 17,7% με εθνικές διαφορές οι οποίες ε, κυμαίνουν ανάμεσα στο 2,4% σε 30,3%. Να μειώσουμε λοιπόν αυτό που μπορεί να θεωρηθεί ως ε, μια πραγματική άβυσος θα πρέπει να αποτελεί μια, μια μόνιμη ε, εργασία μας. Δεν θα πρέπει λοιπόν να παραμείνουν αυτές οι οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες, να επιτύχουμε την πλήρη ένταξη των γυναικών στον κόσμο της εργασίας. Όλα αυτά λοιπόν περνούν μέσα από δράσεις συντονισμένες σε εθνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Χρειάζεται πρώτα απ' όλα να προαγάγουμε όλα τα μέτρα που συμβάλλουν σε μια καλύτερη ε, ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική ζωή και την οικογενειακή ζωή και επίσης να καταπολεμήσουν, να ξεπεράσουμε όλα τα εμπόδια που υπάρχουν για την ένταξη των γυναικών στην οικονομική ζωή. Τον περασμένο μήνα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκ νέου ζήτησε μέτρα απτά να ληφθούν στον τομέα αυτών. Θα πρέπει επίσης τα κράτη-μέλη και οι κοινωνικοί εταίροι να ευνοήσουν μια πιο ισόρροπη συμμετοχή των γυναικών ε, Θέσει υψηλή ευθύνη τόσο στον δημόσιο τομέα όσο και στον ιδιωτικό. Όλα τα αιτήματά μα, όλε οι δράσεις μας, όλα τα αποτελέσματά μας θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο μιας ανακοίνωση που θα φτάσει στον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό πολιτών και δι των γυναικών. Αυτό είναι ο λόγος λοιπόν για τον οποίο στο τρίτο τμήμα της ε, συναντήσεώ μας ε, θα μας ε, παρουσιαστεί αυτό που μπορούν να είναι οι εκστρατείες καταπολέμηση κατά των μισολογικών ανισοτήτων και τον συμβιβασμό ανάμεσα στην οικογενειακή και επαγγελματική ζωή. Χρειάζεται λοιπόν να εμπνευστούμε από αυτού του μηχανισμού για, για, να επικοινωνούμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση και σε επίπεδο κρατών μελών. Εάν το 2014 οι προσπάθειέ μα ε, καρποφορήσουν, τότε οι γυναίκε θα έχουν μια άποψη πολύ πιο σαφή, πολύ πιο θετική για την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα κινητοποιηθούν περισσότερο για τις επόμενες ευρωπαϊκές εκλογές. Τότε θα έχουμε κερδίσει έναν μεγάλο αγώνα ε, ανθρώπινο αλλά και πολιτικό για τη σύγχρονη κοινωνία και για το μέλλον της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ. Quand la présentation commence, Θα αρχίσει παρουσίαση. Παρακαλώ να χαμηλώσετε τα φώτα για να δούμε καλύτερα την οδόνη. Θα καθίσω εδώ για να με βλέπετε και εμένα και τις διαφάνειες, να μην χρειάζεται δηλαδή να μοιράζετε την προσοχή σας. Νομίζω ότι το πρώτο που θα έπρεπε να πω είναι ότι από ό,τι βλέπω μάλλον είμαι ο μόνος ομιλητής ε, σήμερα το απόγευμα, οπότε ελπίζω να δείξετε υπομονή. Θα ήθελα να σας ε, ευχαριστήσω ε, την ομάδα του συναδέλφου. Νομίζω ότι η ομάδα του Τζακ και η δική μου ομάδα συνεργάστηκαν πολύ καλά για ένα πολύ ενδιαφέρον ταξίδι, το οποίο κάνουμε εδώ και δύο χρόνια περίπου. Και τα στοιχεία που θα σας παρουσιάσω σήμερα το απόγευμα είναι και ποσοτικά και ε, ποιοτικά και μέσω του flash, ε, των flash εκτιμήσεων του Ευρωβαρομέτρου και γενικότερα όλων των ε, Διακόπτη Πρόεδρος, θα ήθελα να δώσω το λόγο στην συνάδελφο, την κυρία Κοχμερίν, την Αντιπρόεδρο του Κοινοβουλίου η οποία είναι πρόεδρος της ομάδας υψηλού επίπεδου ε, ισότητας των ευκαιριών ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να ε, σας πω να πάρετε τη θέση σας εδώ, στο βάθρο δίπλα μου, για να είμαστε μαζί, να είμαστε συμπρόεδροι. Ευχαριστώ. Αγαπητές κυρίες και κύριοι, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι για μένα είναι πάντοτε πολύ μεγάλη χαρά να έπομε τη Ρόδης Κράτσα διότι εδώ θα αναλάβω την Προεδρία ε, στο συνέδριο για ε, την ισότητα των φύλων και ε, είμαι πολύ ευτυχής που αναλαμβάνω τη θέση που είχε έως τώρα. Δεν θέλω όμως να καθυστερήσουμε παραπάνω εφόσον έχει ήδη ξεκινήσει η παρουσίαση και στο τέλος μετά την παρουσίαση θα κάνω ορισμένες παρατηρήσεις επί του θέματος που μας απασχολεί σήμερα και ελπίζω ότι στη συνέχεια θα μπορέσουμε να έχουμε μία ενεργητική ε, συζήτηση σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Πρόθεσή μου λοιπόν ε, είναι να προσπαθήσω εντός 20 λεπτών να προσπαθήσω να σας παρουσιάσω τη σύνοψη ε, ενός τεράστιου όγκου δεδομένων που έχουμε στη διάθεσή μας, γιατί όπως και ανέφερα προηγουμένως έχουμε δεδομένα και από τις ε, ειδικέ και από τις συνηθισμένες εκτιμήσεις του Ευρωβαρομέτρου για τα τελευταία δύο με δυόμιση χρόνια. επομένω η πρόκληση για μένα σήμερα είναι να προσπαθήσω να τα συνοψίσω όλα αυτά και να τα αποκρισταλώσω σε μια ε, ιστορία που θα παρουσιάζει μια συνοχή και θα προσπαθήσω να το κάνω. Υπάρχει μια εκτεταμένη εκδοχή της ε, παρουσίαση που θα σας κάνω στο φάκελό σα. Συμπεριλαμβάνονται εκεί όλα τα δεδομένα που θα σα αναφέρω και ορισμένα ε, στοιχεία για το ιστορικό της όλης προσπάθειας, ε, στα οποία θα σας αναφερθώ επίσης. Η, παρουσίασή μου έχει δύο σκέλη σε γενικές γραμμές. Το πρώτο σκέλος αφορά τις σχέσεις μεταξύ των γυναικών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως βασίζεται στα δεδομένα των ε, ερευνών που έχουμε στη διάθεσή μας. Πέντε θέματα να θέσω λίγο το πλαίσιο. Μιλάμε γενικά για την γυναίκα στο πλαίσιο της κοινωνίας. Μετά περνάμε στο θέμα της ανισότητας των φύλων και μετά ε, βλέπουμε πώς έχουν τα πράγματα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μετά περνάμε στις γυναίκες και την πολιτική, τις γυναίκες και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τέλος γυναίκες και οι τελευταίες ευρωεκλογές. Και θα ήθελα σε αυτό το σημείο να κάνω κάποια γενικά, ε, να βγάλω κάποια γενικά συμπεράσματα τα οποία αφορούν ε, την πρόκληση για την οποία ε, ακούσαμε τι ακριβώς θα κάνουμε για να προσεγγίσουμε την ε, πρόκληση αυτή, αλλά βέβαια αυτό θα το αφήσω σε άλλους ομιλητές τουλάχιστον. Θα ήθελα όμως να θέσω την πρόκληση ε, σε σχέση με την έρευνά μας ε, και σε σχέση με τα στοιχεία τα οποία θα εντοπίσω. Είναι πολύ σημαντικό πριν ξεκινήσουμε να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει βεβαίως ένα χάσμα μεταξύ των φύλων, υπάρχουν διαφορές μεταξύ του τρόπου με τον οποίων βλέπουν οι άντρες και οι γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν ε, υπάρχουν τεράστιες διαφορές ε, σε κάθε τομέα. Υπάρχουν σημαντικοί τομείς στους οποίους υπάρχουν διαφορές που πρέπει να αμβληνθούν. Αυτό λοιπόν που θα ήθελα να κάνω είναι απλώς να σας δώσω μερικές ε, πληροφορίες σε σχέση με τη σχέση των γυναικών με την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ήθελα να ξεκινήσω με τις γυναίκες και την ε, κοινωνία. Ακούσαμε ήδη ε, τα δεδομένα που αφορούσαν τα επίπεδα απασχόλησης. Έχουμε τη διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών, 13,7% ε, διαφορά μεταξύ των γυναικών που απασχολούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και των ανδρών. Και αν προσθέσουμε σε, αυτά αυτό το στοιχείο ότι υπάρχουν και γυναίκες που έχουν έχουν προσωρινή απασχόληση σε μεγαλύτερο ποσοστό από τους άνδρες, ότι επίσης δουλεύουν, ε, ασχολούνται με οικιακά στο σπίτι, ε, καταλαβαίνουμε ότι η οικονομική έλλειψη σταθερότητας των γυναικών ε, είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τον ανδρών. Αν δούμε επίσης τους μισθούς, βλέπουμε ότι η διαφορά των μισθών είναι ακόμη μεγάλη. 17,6% λιγότερο είναι σε γενικές γραμμές ε, ε, η διαφορά μεταξύ των μισθών ανδρών και γυναικών και σε μερικές χώρες είναι και άνω του 30%. Χωρίς λοιπόν να θέλω να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες, ε, βλέπετε ήδη ότι υπάρχει χαμηλότερο επίπεδο οικονομικής βεβαιότητας μεταξύ των γυναικών σε σχέση με τους άνδρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη συνέχεια θα ήθελα να μιλήσω για την ισότητα ή ανισότητα των φίλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρώτο που θα ήθελα να πω είναι ότι όταν ε, τους γίνεται ερώτηση, 32% των Ευρωπαίων γυναικών λένε ότι θεωρούν ότι έχουν τύχει άνηση μεταχείρισης σε κάποια χρονική στιγμή, απλώς και μόνο επειδή είναι γυναίκες. Δηλαδή, μία στις τρεις γυναίκες αισθάνονται ότι υπάρχουν ανισότητα σε κάποια πτυχή της ζωής τους και σε κάποια δεδομένη χρονική στιγμή. Αν δούμε τα ε, θέματα για τα οποία θα έπρεπε να δραστηριοποιηθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά την άποψη των γυναικών, βλέπουμε για παράδειγμα το κόκκινο που είναι η άποψη των γυναικών και το μπλε που είναι των ανδρών, του ρωτήσαμε ποιε πρέπει να είναι οι προτεραιότητε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πάνω από το 1 τρίτο των γυναικών είπαν ότι το θέμα τη αντιμετώπιση τη ανισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι ένα από τα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Είναι μια πολύ σαφή απάντηση και είναι και μεγαλύτερο το ποσοστό των γυναικών που το λένε αυτό σε σχέση με τους άντρες ε, και μπορεί να ασχολούνται ε, λιγότερο με ζητήματα όπως ε, για παράδειγμα η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων φτωχότερων χωρών του κόσμου για παράδειγμα. Υπάρχει λοιπόν μια διαφορά εστίασης μεταξύ ανδρών και γυναικών σε σχέση με τις προτεραιότητες που θα ήθελαν να δουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, θέτει. Τώρα, όσον αφορά το θέμα των γυναικών και της πολιτικής, έχουμε κάποια δεδομένα για την αναλογία των γυναικών που ο κόσμος θα ήθελε να υπάρχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 48% ε, μας είπαν ότι θα ήθελαν 50% τουλάχιστον των ε, γυναικών, των ευρωβουλευτών να είναι γυναίκες ε, και βλέπουμε επίσης ότι και οι γυναίκες θα ήθελαν να συμμετέχει σε σημαντικό βαθμό, να είναι δηλαδή σημαντικότερο το ποσοστό των γυναικών ευρωβουλευτών. 34% ε, είναι ήδη ε, γυναίκες ε, ευρωβουλευτές και όπως βλέπετε συνεπώς υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Νομίζω ότι τώρα, μετά το γυναίκες και πολιτική, πλησιάζουμε περισσότερο στο επίκεντρο της σχέσης μεταξύ των... της σχέσης γυναικών και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα ερώτημα που θα έπρεπε να θέσω πριν αναφερθούμε στη σχέση των γυναικών με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ευρωεκλογέ είναι η σχέση των γυναικών με την πολιτική γενικώ. Πόσο δηλαδή ε, συμμετέχουν και νομίζω ότι όταν ρωτάει κανείς τον κόσμο, όταν ας πούμε συναντιέται με τους φίλους του, συζητάτε τα πολιτικά ή όχι, οι γυναίκες έχουν την τάση να λένε ότι δεν συζητούν ποτέ πολιτική κατάσταση με, με, με τους φίλους τους, ε, ότι συνήθως αυτή είναι μια κουβέντα που θα κάνουν οι άντρες περισσότερο. Είναι πάντως ενδιαφέρον το ότι οι στατιστικές ε, ε, δείχνουν ότι οι γυναίκες ασχολούνται λιγότερο με την πολιτική. Όταν λοιπόν μιλούμε για την πολιτική και ειδικότερα για ε, τα στοιχεία εστίασης της πολιτικής, οι γυναίκες έχουν διαφορετικά σημεία εστίασης από τους άντρες. Για παράδειγμα, ποια είναι η πολιτική εστίαση, αν κάνουμε αυτή την ερώτηση και δούμε τα δεδομένα, είτε πρόκειται εθνικό, για εθνικό, τοπικό, περιφερειακό ή ευρωπαϊκό επίπεδο, οι γυναίκες ε, κατά, σε, κατά, ε, ε, κατά μεγαλύτερο ποσοστό ε, το τοπικό και περιφερειακό επίπεδο είναι πιο σημαντικό για τις γυναίκες από ότι για τους άντρες ενώ οι άντρες θεωρούν ότι το εθνικό και το ευρωπαϊκό επίπεδο είναι αυτό που επηρεάζουν περισσότερο τη ζωή τους. Είναι επίση ενδιαφέρον ότι υπάρχουν πολύ σαφείς απόψεις που ακούσαμε από την πρόσφατη ποιοτική μελέτη που έγινε και θα σας ε, διαβάσω μερικά από αυτά. Για παράδειγμα, μια χώρα στην Ολλανδία είπε ότι εγώ θα προτιμούσα να επενδύσω προσπάθειες σε τοπικό επίπεδο, γνωρίζω καλύτερα τον κόσμο, τα κίνητρα είναι μεγαλύτερα. Υπάρχει λοιπόν κάτι, για την, κάτι που έχει σχέση με την εγκύτητα. Κάποια από τη Σλοβακία μας είπε «Εγώ παθητικά παρακολουθώ και όταν μου ζητούν να πω την άποψή μου, τι λέω. Συνήθως ασχολούμαι όμως με πράγματα που επηρεάζουν εμένα και την οικογένειά μου». Και βλέπετε και δύο ακόμη ε, παραθέσεις. Κάποιος είπε δεν με ενδιαφέρουν όλα αυτά, είναι πολύ μακριά από μένα. Με ενδιαφέρει να ασχολούμαι με πράγματα ε, που, απασχολούν, που επηρεάζουν την καθημερινή μου ζωή και για τα οποία πιστεύω ότι η άποψή μου επηρεάζει την πραγματική μου ζωή. Και επίση, ναι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ναι, υπάρχει, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να έχει τον αντίκτυπο μια πραγματικής κυβέρνησης. Όλες αυτές οι παραθέσεις δείχνουν ότι οι γυναίκε έχουν την τάση να ενδιαφέρονται και να επηρεάζονται περισσότερο από πράγματα που έχουν να κάνουν με τη ζωή του, με την οικογένειά τους, με πιο απτά πράγματα καθημερινά, σε σχέση με, τον, με τους άντρες οι οποίοι βλέπουν την ευρύτερη εικόνα και πέρα από την δική τους ζωή. Αυτή είναι λοιπόν μια εικόνα που υπάρχει γενικά. Τώρα, ποιοι είναι οι τομεί που ενδιαφέρουν τις γυναίκες και όπως ενδεχομένως να περιμένει κανείς, ε, είναι τα ζητήματα που επηρεάζουν πιο άμεσα την καθημερινή ζωή, ε, τη δική τους, των οικογενειών τους και των κοινοτήτων στις οποίες ανήκουν. Για παράδειγμα, βλέπετε η αύξηση των τιμών και ο πληθωρισμός ε, 3% ε, περισσότερες γυναίκες ε, ανησυχούν για αυτό το ζήτημα, ε, ενώ για την οικονομική κατάσταση γενικότερα 5% λιγότερο οι γυναίκες ασχολούνται γι' αυτό. Όπως επίσης τα θέματα της σύνταξης, όλα αυτά θα θεωρούν οι γυναίκες πιο απτά ζητήματα σε σχέση με τους άντρες. Κάτι ακόμη για τα ζητήματα τα οποία θα ήθελα να δουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αντιμετωπίζει. Ορισμένες πολιτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο θεωρούν ότι η εξωτερική πολιτική πρέπει να έχει ε, μεγαλύτερη ε, σημασία το θέμα της ε, πολιτικής των καταναλωτών. Για παράδειγμα, κατά 4% πιστεύουν οι γυναίκες ότι πρέπει να είναι σημαντικότερο ε, σε σχέση με τους άντρες. Το θέμα ε, το φορολογικό, η κοινή ενεργειακή πολιτική είναι πιο κάτω στις προτεραιότητες. Η καταπολέμηση όμως της τρομοκρατίας, του σεβασμού του, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, αυτά είναι ένα, αυτά είναι, αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα για τις γυναίκες ε, οι γυναίκες δηλαδή έχουν μια ε, πιο κοινωνική ατζέντα θα λέγαμε σε σχέση με πολιτική, οικονομική ατζέντα, ατζέντα σε μακροοικονομικό επίπεδο. Τώρα, σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ποια είναι η σχέση των γυναικών με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μία απλή ερώτηση. Πόσο πιστεύουν ότι γνωρίζουν οι γυναίκες για την Ευρωπαϊκή Ένωση, πόσα πιστεύουν ότι γνωρίζουν. Συμφωνείτε ή μάλλον διαφωνείτε ε, ότι γνωρίζετε πώς δουλεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 12% λιγότερο οι γυναίκες σε σχέση με τις γυναίκες, 51% δηλαδή ε, οι άντρες ε, και 39% ε, οι γυναίκες ε, θεωρούν ότι μάλλον θα έπρεπε να διαφωνήσουν με, το, με την απλή πρόταση δεν γνωρίζω αρκετά για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 77% των γυναικών λένε ότι δεν είναι καλά ενημερωμένες για τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έναντι 69% των ανδρών. 69 με 77 είναι αρκετά μεγάλη διαφορά. Γνωρίζουν λοιπόν λιγότερο καλά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποια όμω είναι η άποψή του για την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα αναφερθώ σε κάποια στατικά στοιχεία που ακούσαμε και προηγουμένω. Έχουμε διάφορε μετρήσει. Έχουμε την εικόνα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ποια είναι γενική. Και αν δει, για παράδειγμα, κανεί το πράσινο κομμάτι του ε, γραφήματο, ε, αυτέ είναι οι θετικέ απαντήσει σε σχέση με την εικόνα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, με την ε, αξία της, του γεγονότος ότι η χώρα μου ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σε κάθε περίπτωση βλέπουμε ότι Συγγνώμη, ε, τα έχουμε βάλει ανάποδα Όπου γράφει γυναίκε, ε, θα έπρεπε να γράφει άντρε και το αντίστροφο. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα εδώ με την παρουσίασή μου. Ζητώ συγγνώμη, αλλά εν πάση περιπτώσει η πραγματικότητα είναι ότι το πράσινο αφορά του άντρε. 51% έχουν μια θετική γενική εικόνα ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 45% οι γυναίκε. 57% ε, των ανδρών θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι καλό πράγμα για τη χώρα του. 48% των ανδρών σε σχέση με 46% των γυναικών ε, εμπιστεύονται την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν λοιπόν μεγάλες διαφορές όπου ε, διαφαίνεται μια σαφή στάση όπως βλέπετε. Και αν δούμε και συγκεκριμένες ευρωπαϊκές πολιτικές όπως για παράδειγμα την νομισματική ε, ένωση. 65% των ανδρών είναι υπέρ του ενιαίου νομίσματος και της νομισματικής ένωσης ενώ 57% είναι οι γυναίκες. 73% των ανδρών ε, είναι υπέρ της κοινή εξωτερικής πολιτικής ε, σε σχέση με 65% των γυναικών. Το ίδιο θα ίσχυε και για την ε, κοινή εξωτερική πολιτική και για την πολιτική της διεύρυνσης. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις οι γυναίκες παρουσιάζουν χαμηλότερα ποσοστά από τους άντρες. Υπάρχουν όμως και τομείς τους οποίους, όπως είπα και προηγουμένως, ε, θεωρούν γυναίκες ότι θα έπρεπε να κάνει περισσότερη η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως για παράδειγμα βελτίωση της προστασίας του καταναλωτή, της δημόσιας υγείας, 39% ε, γυναίκες, 33% άνδρες, ε, καταπολέμηση τρομοκρατία, σεβασμός της προσωπικής ελευθερίας, περισσότερα, μεγαλύτερα ποσοστά οι γυναίκες από τους άντρες. Ε, όπως βλέπετε, ε, προς τα κάτω, η ενεργειακή πολιτική, η πολιτική ασφάλειας, για παράδειγμα, δεν είναι πολιτικές που είναι στην προτεραιότητα των γυναικών, γιατί κυρίως κοινωνικά θέματα είναι αυτά που απασχολούν τις γυναίκες, όπως φαίνεται μία ακόμη φορά. Όπως είπα και στο προηγούμενο τμήμα της παρουσίασής μου, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Θέλουν λοιπόν οι γυναίκες ε, μια κοινωνική ατζέντα ακούσαμε ήδη ότι έχουν λιγότερο θετική άποψη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και άμα τους ρωτήσουμε θεωρείτε ότι το συμφέρον σας ως γυναίκας εκπροσωπείται καλά από την Ευρωπαϊκή Ένωση 46% το κόκκινο και το πορτοκαλί μαζί λένε όχι, όχι, όχι ιδιαίτερα ενώ 39% θεωρούν ότι, ότι το, τα συμφέροντά τους εκπροσωπούνται σχετικά καλά ή καλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά, αυτά είναι λοιπόν τα στοιχεία ε, βάσει των οποίων κλήθηκαν να ψηφίσουν οι γυναίκες στις τελευταίες ευρωεκλογές. Και να δούμε λοιπόν αυτά με περισσότερη λεπτομέρεια. Το επίπεδο ενδιαφέροντος ε, σε ευρωεκλογέ 55% των ε, γυναικών είπαν ότι δεν ενδιαφέρονται ή δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τις ευρωεκλογέ ε, σε σχέση με 48% ε, των ε, ανδρών. Εντάξει, δεν είναι μεγάλη έκπληξη σε σχέση με αυτά που ακούσαμε ως τώρα. Αλλά νομίζω ότι είναι αρκετά συνεπή τα πράγματα ε, όσο συνεχίζουν τα διάφορα στατιστικά στοιχεία, αλλά όπως είπα και προηγουμένως, η διαφορά στην ψηφοφορία δεν φάνηκε να αντικατοπτρίζει τις προσδοκίες μας, δηλαδή διαφορά μεταξύ 8 και 10 ποσοστιαίων μονάδων. Όμως, μόνο 2% λιγότερες ήταν οι γυναίκες που ψήφισαν σε σχέση με τους άντρε. Σε μερικές χώρες ε, όχι μόνο ήταν πολύ κοντά τα ποσοστά, αλλά υπήρχαν και χώρες τις οποίες οι γυναίκες προσήλθαν περισσότερο στις κάλπες από ότι οι άνδρες. Έχουμε λοιπόν δεδομένα ε, για το γιατί ψήφισε κάποιος, ρωτήσαμε και άνδρες και γυναίκες γιατί ψηφίσετε και οι ερωτήσεις, ε, οι απαντήσεις που ακούσαμε ήταν σε μερικές φορέ παρόμοιε. Είναι το καθήκον μου ω πολίτη για παράδειγμα. Οι γυναίκες συνήθως ε, πιο εύκολα το λένε αυτό από ότι οι άντρε ή ας πούμε είμαι υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λιγότερες γυναίκες έδωσαν αυτό ως λόγο. Αλλά βέβαια αυτό δεν εξηγεί όλη την κατάσταση. Ποια είναι τα ζητήματα που οδήγησαν τις γυναίκες στο να ψηφίσουν. Η ανεργία, το μέλλον των συντάξεων, η ασφάλεια των τροφίμων, όλα αυτά είναι τα ζητήματα που οδήγησαν τις γυναίκες να ψηφίσουν, ενώ η οικονομική ανάπτυξη, ας πούμε, δεν ήταν παράγον που τις οδήγησε στις κάλπες. Δεν υπάρχει λοιπόν ένας παράγοντας, υπάρχει ένας συνδυασμός παραγόντων. Τώρα, για αυτές που δεν ψήφισαν, γιατί δεν ψήφισαν. Μπορούμε να, συγκρίνουμε τι είπαν, να συγκρίνουμε τι είπαν οι άντρες και τι είπαν οι γυναίκες. Για παράδειγμα, ο παράγοντας της, ε, του μη ενδιαφέροντος για την πολιτική. δεν γνωρίζω πολλά για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό ε, δεν ψήφισα. Αυτό το λένε πολύ περισσότερο οι γυναίκες από ότι οι άντρες. Τι συμβαίνει, αναρωτηθήκαμε. Γιατί οι γυναίκες ασχολούνται λιγότερο με την Ευρωπαϊκή Ένωση από ότι άντρε. Δεν είναι απλή απάντηση. Προσπαθήσαμε με τα δεδομένα που σα παρουσίασα και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που είχαμε στη διάθεσή μα να κάνουμε μια υπόθεση. Κάπω έτσι έχουν τα πράγματα, όπω φαίνεται στη διαφάνεια. Δεν είναι ένα παράγον, είναι διάφοροι παράγοντε που συνδέονται μεταξύ του, αλλά ο τρόπο με τον οποίο ε, αλληλεπιδρούν ο ένα με τον άλλον έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργείται ένας κύκλος ο οποίος οδηγεί στην ενίσχυση αυτής της αίσθησης απόστασης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάνω αριστερά, για παράδειγμα. Οι γυναίκες θεωρούν ότι δεν είναι πολύ σχετικοί ε, με εκείνες ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, ενδιαφέρονται λιγότερο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και επειδή ενδιαφέρονται λιγότερο, κάνουν λιγότερη προσπάθεια να μάθουν περισσότερα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, δεν ε, δεν ακούν ε, τόσο πολύ αυτά που τους παρουσιάζουν, για παράδειγμα, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και γι' αυτό το λόγο στη συνέχεια θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι το πιο μακρινό σε σχέση με εκείνε και γι' αυτό θεωρούν βέβαια ότι δεν τι επηρεάζει πολύ. Μπορεί λοιπόν να δημιουργηθεί μια τάση η οποία είναι αυτοτροφοδοτούμενη ουσιαστικά. Ένας φαύλο κύκλο για να το πω έτσι. Εδώ ολοκληρώνεται το πρώτο τμήμα. Κρατήστε αυτήν τη σκέψη. Και το δεύτερο τμήμα θα ήθελα να επανέλθουμε μετά στο τέλος σε αυτό για να σας πω να το ξανασυζητήσουμε. Λοιπόν, πώς αντιμετωπίζουμε τις γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακούσαμε ήδη πολλές στατιστικές ότι βελτιώνεται η κατάσταση όσον αφορά την απασχόληση, το ποσοστό ανεργίας που έχει μειωθεί, ε, η μερική εργασία είναι κάτι το οποίο ακόμη υπάρχει αλλά έχουν γίνει πρόοδοι. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιέζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να υπάρχει ίση αμοιβή τα κράτη-μέρη για να λύσουν το πρόβλημα της ανεργίας των γυναικών. Καταρτίζει η ε, νηπιαγωγία, ιδρύματα να βοηθούν τους ηλικιωμένους, ε, κινητοποιεί για μεγαλύτερη ανάληψη ευθύνης. Όλα αυτά τα ακούσαμε. Ακούσαμε επίσης ότι έχει ευξηθεί και ο αριθμός των γυναικών ευρωβουλευτών τα τελευταία χρόνια και είναι πολύ καλύτερη η κατάσταση από ό,τι στα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών. Μιλήσαμε επίσης για τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν στις ευρωεκλογές, την ανεργία, την αμοιβή. Ε, γνωρίζουν ότι θέλουμε περισσότερες πληροφορίες σαν τα δικαιώματά τους ως πολίτες, τα μέτρα για την εκπαίδευση, για την ε, πολιτική συνεργασία. Βλέπουμε λοιπόν ότι το Κοινοβούλιο ε, κάνει αυτά τα οποία θέλουν οι γυναίκες τα οποία θα μπορέσουν να λύσουν ε, τα προβλήματα αλλά κατά κάποιον τρόπο αυτά τα θέματα δεν ανακοινώνονται γιατί οι γυναίκες βρίσκονται σε ένα φαύλο κύκλο ο οποίος ενισχύεται όσο περνάει ο χρόνος. Άρα το, η πρόκληση είναι πώς αυτός ο φαύλος κύκλος θα σπάσει. Διότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να ε, κουνούμε απλώ το δάχτυλο και να ζητούμε κάτι άλλο. Μπορούμε να προσπαθήσουμε να τους μιλήσουμε, να τους εκπαιδεύσουμε. Αλλά εάν κάποιος δεν σε ακούει δεν μπορεί να περάσει το μήνυμα. Ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση βέβαια μπορείτε να ε, χοροπηδάτε και να λέτε εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Αλλά αυτό δεν λύνει το πρόβλημα. Ε, τα θέματα όμως της Ευρωπαϊκής Ενώσεως απασχολούν όλες τις γυναίκες ε, και ε, εμείς θεωρούμε ότι ίσως ε, εδώ σε αυτό το σημείο μπορούμε να σπάσουμε το φαυλοκύκλο και αν σπάσουμε το φαυλοκύκλο αν πείσουμε τις γυναίκες ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σημασία αναγνωρίζει τα προβλήματά τους θα προσελκυθούν θα ενδιαφερθούν περισσότερο θα γνωρίσουν καλύτερα την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο γνωρίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πλησιάζουν και όσο πλησιάζουν θα πιστούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σημασία για αυτές. Ε, βέβαια ίσως είναι προφανές να το λέω εγώ σαν ερευνητής αλλά θα πρέπει άλλοι να αποφασίσουν πώς θα μπορέσουμε να σπάσουμε αυτό το φαύλο κύκλο και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση, η οποία εν μέρη παρουσίασε τρομακτικούς αριθμούς. Διότι ε, βλέπουμε ναι μεν περισσότερες γυναίκες στο Ευρωκοινοβούλιο και ε, ιδίω ε, θεωρώ ότι οι γυναίκες θεωρούν ότι εμπλέκονται στην διαδικασία της Ευρώπης και ελπίζουμε ότι στα επόμενα έτη θα μπορέσουν καλύτερα να οδηγήσουν σε ένα πιο θετικό αποτέλεσμα ε, είτε από συμμετοχή ψηφοφόρων γυναικών είτε εκλεγμένων γυναικών. Παρ' όλα αυτά όμως θα έπρεπε να πούμε κάτι το οποίο είναι πάντοτε δύσκολο. Δηλαδή υπάρχουν τώρα πολλά στοιχεία τα οποία ε, αναφέρονται και ισχύουν για όλες τις Ευρωπαίες όπως είπατε και εσείς. αυτά όμως αν θέλουμε να επέμβουμε πολιτικά και να δούμε τι ε, πρόοδος μπορεί να γίνει θα σας έλεγα ότι καλύτερα θα ήταν να ξεκινήσει η συζήτησή μας αμέσως εσείς μπορείτε να μας πείτε τις εμπειρίες σας, τις προτάσεις σας για το πως μπορεί κανείς να πλησιάσει καλύτερα τις γυναίκες και να τις προσελκύσει στα ευρωπαϊκά τεκτενόμενα και να κάνουμε μια επικοδομητική συζήτηση. Καλύτερα να μιλήσω αγγλικά. Είμαι πρώην Ευρωβουλευτήνα και μέλος της Επιτροπής Γυναικών. Ε, ήμουνα εδώ επί τρεις και συμμετείχα σε όλες τους προεκλογικούς αγώνες, ιδίως προσπαθώντας να προσεγγίσω τις γυναίκες. Όσον αφορά την επικοινωνία και το συζητήσαμε ήδη αυτό με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η επικοινωνία λέγω αυτή δεν γίνεται βάση της προτεραιότητας των γυναικών, δεν αναφέρεται εις τις πτυχές της ζωής των γυναικών και ένας άλλος λόγος είναι ότι βεβαίως οι κυβερνήσεις των κρατών μελών όποτε υπάρχουν δυσάρεστα νέα τα οποία πρέπει να αναφερθούν τα βάζουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση Ξέρετε, ε, μιλήσατε γερμανικά και τη Γερμανία και την Αυστρία λένε όιρο τόιρο, δηλαδή το ευρώ ακριβένει και ανεβαίνει το κόστος ζωής και ξέρετε ότι παρόλο που έχουν μειωθεί πολλές τιμές βασικών πρώτων υλών αυτό ισχύει. Άρα η Επιτροπή Γυναικών θα έπρεπε να εξετάσει το θέμα αυτό, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσει να επικοινωνήσει. Ε, να δούμε τι τύπο διαβάζουν οι γυναίκες πώς τοποθετούνται για να μπορέσουμε να καλέσουμε τις γυναίκες ε, δημοσιογράφους παραδείγματος χάρη σε ορισμένες ακροάσεις διότι πριν από μερικές εβδομάδες έγινε ένα σεμινάριο σχετικά με το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση για την βία εναντίον των γυναικών και το πρόβλημα του βιασμού σαν έγκλημα πολέμου. Θυμάμαι ότι την εποχή του πολέμου στη Βοσνία είχε οργανωθεί η ε, σχετική ακρόαση και οι γυναίκες ήταν πάρα πολύ ευαίσθητες. Αυτά όμως ε, μείνανε και τα αποτελέσματα και κλεισμένων των θυρών. Και η Μαντλέν Ολμπράιτ μου είχε ζητήσει να επαναφέρω το θέμα επιτάπητος και η Επιτροπή, στην Επιτροπή Ελευθεριών στην Επιτροπή Γυναικών νομίζω υπάρχει ένα ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τον βιασμό το οποίο ανέρχεται σε δύο χρόνια και το οποίο πρέπει να το στηρίξουμε στον ΟΗΕ. Ε, θα έχουμε την έκθεση του Πεκίνου 15 χρόνια μετά. Ε, όλα τα θέματα τα οποία είχαν συζητηθεί στο Πεκίνο πριν πριν 15 χρόνια, δέστε τα, δούμε τι έχει γίνει και να δούμε πώς θα εμπλέξουμε τον τύπο που ε, απευθύνεται στις γυναίκες και δεν αναφέρουμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Le Monde, όχι αναγκαία. Ευχαριστώ. σε ε, μία τελευταία συνεδρίαση του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, συζητήσαμε πώς ε, θα οργανώσουμε τον εορτασμό της 9ης Μαΐου και η ιδέα ήταν να γίνει ένα αγώνας ποδοσφαίρου και ορισμένες γυναίκες είπαν ότι αυτό θα ήταν ίσως πιο ενδιαφέρον για τους άντρες από ότι για τις γυναίκες και αν θέλετε να προσελκύσετε γυναίκες απολυτικά δηλαδή ανεξάρτητα της πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό που θα ήταν καλό θα ήταν να γίνουν ορισμένα πράγματα τα οποία να ενδιαφέρουν κατά προτεραιότητα και τις γυναίκες να μην υπάρχει δηλαδή διαχωρισμός το, το βόλεϊ παραδείγματος χάρη τουλάχιστον το ποδόσφαιρο είναι πολύ καλό για τις γυναίκες ποδοσφαιριστές στη Γερμανία που είναι πιο επιτυχής και από τους ε, άντρες και είναι διεθνούς επίπεδου αλλά όσον αφορά το γενικότερο ενδιαφέρον νομίζω ότι είναι μπουσιώδες και θα έπρεπε να βρούμε κάποιον άλλον τρόπο να δούμε πώς θα το προωθήσουμε. Το όνομά μου είναι Καρίνα Ροτ. Ήμουνα επικεφαλής της Σχετικής Επιτροπής στο ε, ε, το ε, Συμβούλιο της Ευρώπης και σε ένα μεγάλο λόμπι για τις γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το οποίο με ενοχλεί στην έκθεση αυτή κατά κάποιον τρόπο και συγχρόνως με προσέλκυσε είναι ότι οι γυναίκες θα ήθελαν να έχουν περισσότερους βουλευτές και ευρωβουλευτές και παρόλα αυτά όταν υπάρχουν οι ευρωεκλογέ δεν έχετε περισσότερες γυναίκες υποψήφιες και είναι κάτι περίεργο το οποίο δεν αναφέρεται ότι εξαρτώμαστε από τα πολιτικά κόμματα και ε, ε, αυτοί καθορίζουν ποιος θα συμμετάσχει, ε, θα συμμετάσχει στις επιτροπές και αν αυτοί δεν προτείνουν γυναίκες πώς θα έχουμε υποψηφίους. Είναι πολύ απλό αλλά κανείς δεν το αναφέρει και γι' αυτό ήθελα εδώ να το τονίσω. Δεν νομίζω ότι αν οι γυναίκες δεν ψηφίζουν, δεν ενδιαφέρονται για την Ευρωπαϊκή Ένωση Πιστεύω ότι το θέμα που τους ενδιαφέρει πάνω απ' όλα είναι ε, το θέμα που δεν έχει αλλάξει τίποτα παρόλο που έχουμε πολλές αλλαγές από το 57 και τη συνθήκη της Ρώμης αλλά τα ουσιαστικά θέματα των γυναικών ακόμη δεν έχουν επιληθεί. Το οικονομικό, διότι όπως είπατε υπάρχει ένα κενό όσον αφορά την αμοιβή. Δεν ε, βρίσκονται στα διοικητικά συμβούλια σε ορισμένες ε, χώρες ε, γίνεται μία προσπάθεια για τις γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια παρόλα αυτά όμως δεν είναι ικανοποιητικό το αποτέλεσμα και βλέπετε ότι οι γυναίκες είναι σαν να μην υπάρχουν. Όταν λοιπόν κοιτάξτε ε, τους ε, κανόνες οικονομικών οι περισσότεροι καταρτίζονται από άντρες και επηρεάζουν τη ζωή των γυναικών και υπάρχει η υπουργό Οικονομικών στη Γαλλία γυναίκα αλλά στις περισσότερες άλλες χώρες δεν ισχύει αυτό. Μετά, η βία. Η βία είναι πάρα πολύ υψηλή, είτε πρόκειται για την οικογενειακή βία, για την πορνεία, για τους υποχρεωτικούς γάμους. Είναι θέματα με τα οποία θα έπρεπε να ασχοληθούν οι γυναίκες και δεν ασχολούνται. Και όπως ε, είπε και η κυρία για τα Βαλκάνια και το έγκλημα πολέμου, υπάρχει και κάτι ακόμη. Υπάρχει η εμπορία ε, το, ε, ε, ανθρώπων και όπως είπα δεν λαμβάνουν οι γυναίκες αρκετές αποφάσεις στη δημόσια ζωή. Δεν βλέπουμε στην κορυφή της Ευρώπης τόσες γυναίκες τώρα. Όταν έχουμε υποψηφίους για τις ε, ύψιστες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι γυναίκες δεν υπήρχαν καθόλου. Δεν παρουσιαζόντουσαν. Όσο λοιπόν οι γυναίκες βλέπουν ότι υπάρχει κάτι τέτοιο δεν ε, πρόκειται να λυθούν τα προβλήματα, δεν πρόκειται να υπάρχει αξιοπιστία και η κατάσταση απλώς είναι αυτή. Σήμερα το πρωί ήμουν σε ένα ε, ε, ε, σε, μια στρογγυλή τράπεζα στην Λουβάν Λανόβ σχετικά με τη φτώχεια και μου έκανε εντύπωση οι γυναίκες προσπαθούν να επιβιώσουν τις κρίσεις κάθε μέρα η οικονομική κατάσταση των γυναικών αυτών είναι τόσο τραγική στην Ευρώπη οι γυναίκες χάνουν τη δουλειά τους συνέχεια με ένα ρυθμό που δεν μπορείτε καν να φανταστείτε και πρέπει να μεγαλώσουν, να αναθρέψουν τα παιδιά τους μόνες τους. Ορισμένες από τις γυναίκες αυτές, σαν αυτές που είδα σήμερα το πρωί, έλεγαν ότι τόσο ντρέπουμε για την εικόνα που δίνω στα παιδιά μου, διότι η εικόνα μου έχει τόσο καταρρεύσει, αλλά δεν μπορώ να τους προσφέρω τα αναγκαία προς το ζήν και γι' αυτό έχουν μια κακή εικόνα για μένα. Πολλές γυναίκες μιλούσαν για τη βία την οποία υφίστανται από την κοινωνία και την έλλειψη σεβασμού από τις αρχές γιατί είναι φτωχές. το οποίο είναι ακόμη χειρότερο. Με συγχωρείτε που μακρηγόρησα, αλλά για αυτή είναι η λόγη για τους οποίους οι γυναίκες ε, οι οποίες ε, έχουν συγκεκριμένους στόχους αισθάνονται ότι δεν εισακούονται παρκώς. Ευχαριστώ. Προφανώς θέσατε πολλά σημαντικά θέματα όταν ε, αναφερθήκατε ε, στο ρόλο των πολιτικών ομάδων που πρέπει να προωθήσουν τις γυναίκες ένας από τους επόμενους ομιλητές θα αναφερθεί στις γυναίκες υποψηφίους άρα το θέμα αυτό θα παρουσιαστεί και πρέπει να εστιάσουμε τη συζήτηση στο θέμα αυτό αργότερα. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και θα πρέπει σε ορισμένα κράτη-μέρη να μπορεί κανείς να προωθήσει υποψηφίους και πετύχεται το θέμα της ισότητας των φύλων που δεν αντιμετωπίζεται παντού με τον ίδιο τρόπο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ είμαι Ευρωβουλευτής ε, της Πολωνίας και είμαι επίσης ε, μέλος μιας ε, πρωτοβουλίας στην Πολωνία. Πάνω από 100.000 υπογραφές συλλέξαμε και προσπαθούμε να περάσουμε ένα νομοσχέδιο για ποσόστοση των γυναικών στην πολιτική στην Πολωνία. Είπατε ότι η κοινωνική μιλήσατε ότι, είπατε ότι οι γυναίκε ε, ενδιαφέρονται πολύ περισσότερο για την κοινωνική ατζέντα και είπατε, υπονοήσατε ότι αυτό δεν είναι πολιτική ατζέντα Όμω, νομίζω ότι όπω δείχνει και η κυβέρνηση Ομπάμα δεν άσχετα αυτά μεταξύ του. είναι γεγονό ότι κοινωνική ατζέντα προτιμούν οι γυναίκε, αλλά κάνατε μια διαφορά με, κάνατε τη διάκριση με την πολιτική ατζέντα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ασχολείται με κοινωνικά θέματα αλλά ίσως θα έπρεπε να ζητήσουμε από τις γυναίκες να ασχοληθούν ε, και να ενδιαφέρονται ε, και με την πολιτική γενικότερα, όχι μόνο με κοινωνικά θέματα. Οι γυναίκες ε, να μην είναι μόνο στις επιτροπές που ασχολούνται με τα κοινωνικά θέματα, αλλά και στις υπόλοιπες επιτροπές, για παράδειγμα για την υγεία. Οι γυναίκες δεν ε, φαίνονται να ασχολούνται ιδιαίτερα με πιο απτά ζητήματα, ότι όλο και περισσότερο απασχολούνται στους κοινωνικούς τομείς και ίσως θα έπρεπε ακριβώς να τις ενημερώσουμε περισσότερο για περισσότερα πολιτικά θέματα για να μπορέσουν ε, να προσεγγίσουν περισσότερο την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όσον αφορά τις περιφέρειες, δείτε τις περιφερειακές εκλογές. Είπατε ότι ασχολούνται περισσότερο με ζητήματα που είναι πιο κοντινά σε εκείνες. Πολύ περισσότερες γυναίκες συμμετέχουν ε, στις τοπικές, στα τοπικά πολιτικά ζητήματα. Πολύ περισσότερες προσέρχονται στις κάλπες όταν πρόκειται για εκλογές σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο. Όχι, όταν έχουμε 22% προσέλευση στις ευρωεκλογέ, όπως έγινε για παράδειγμα στην Πολωνία και σε άλλες χώρες, ε, δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία αν 2% παραπάνω ήταν οι άντρες από τις γυναίκες. Το θέμα είναι πώς γνωστοποιεί κανείς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλο τον πληθυσμό. Ευχαριστώ πολύ. Λέει η Πρόεδρος, πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης, δηλαδή τα μέσα ενημέρωσης και γυναικείες υποψηφιότητες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η κυρία Στρέλα είναι ήδη εδώ, θα ήθελα να δώσω την δυνατότητα στον πρώτο μας ομιλητή να απαντήσει στα σχόλιά σας. Ναι. Για το τελευταίο αυτό σχόλιο που κάνατε, αν έδωσα την εντύπωση ότι έκανα τη διάκριση ανάμεσα στα κοινωνικά θέματα και την πολιτική, όχι αυτή δεν ήταν καθόλου η πρόθεσή μου. Η πρόθεσή μου ήταν να μιλήσω για το πού εστιάζεται η πολιτική ατζέντα και να μιλήσουμε για ζητήματα ε, τα οποία γίνονται πιο γνωστά και φαίνεται ότι οι γυναίκες... Ε, προσλαμβάνουν καλύτερα τα μηνύματα που αφορούν την ε, δική του ζωή, την οικογενειακή του ζωή και την ε, ευρύτερη ζωή της κοινότητά τους και μερικές φορές λιγότερο ενδιαφέρονται για ζητήματα μακροοικονομικής πολιτικής ας πούμε. Βέβαια αυτές είναι γενικεύσεις, μεγάλες γενικεύσεις, αλλά πιστεύω ότι είναι ζήτημα ε, εστίασης ε, της πολιτικής ε, ατζέντα. Δεν είναι ζήτημα δηλαδή του να λέμε αν το ένα θέμα είναι πολιτική και το άλλο δεν είναι. Νομίζω ότι συμφωνούμε. Απλώς πήρα το λόγο για να πω ότι, για να εξασφαλίσω ότι δεν υπάρχει καμία παρεξήγηση των όσων είπα. Ναι και θα ήθελα να συνεχίσω και εγώ αυτό που είπε ο προλαλή σα το ερώτημα για την ε, νομισματική ένωση, για παράδειγμα, ήταν πολύ ενδεικτικό. Όταν ρωτήθηκαν οι γυναίκες αν συμφωνούν, αν το υποστηρίζουν ή όχι. Τα ζητήματα του προϋπολογισμού, τα ζητήματα του νομίσματος ε, ενδιαφέρουν πολύ περισσότερο τις γυναίκες από ό,τι άλλα. Γι' αυτό οι γυναίκες απάντησαν θετικά σε αυτό το ερώτημα. Αυτό νομίζω ότι δείχνει ακριβώς ε, αυτό που είπε ο Πολ προηγουμένως, ότι αυτά είναι πολιτικά ζητήματα βεβαίως, απλώς ε, πλαισιώνονται με έναν κοινωνικό τρόπο και τότε μόνο οι γυναίκες ανταποκρίνονται καλύτερα και συμμετέχουν περισσότερο. Thank you very much Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας και ευχαριστώ πολύ για τον πρώτο αυτό γύρο συζήτησης. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Εστρέλα για το επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης. to everybody. Καλησπέρα σας. Υπάρχει πορτογαλική διερμηνία, ως εκ τούτου θα συνεχίσω στην μητρική μου, την πορτογαλική. Φτάσαμε στο δεύτερο τμήμα της σημερινής μέσης διατάξεως και θα μιλήσουμε για τα μέσα ενημέρωσης και τις γενικές υποψηφιότητες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα ως εκ τούτου να δώσω κάποιες ιδέες για την συζήτηση που θα ακολουθήσει και στηρίζομαι λίγο πολύ και στις δικές μου εμπειρίες αλλά και στο ζήτημα των ποσοστώσεων σχετικά με τις γυναίκες. Και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ένα κείμενο της Χίλαρη Κλίντον. Ένα κείμενο πρόσφατο, το οποίο αναφέρει ότι σήμερα υπάρχουν περισσότερε γυναίκε στις επιχειρήσει, στις κυβερνήσει και στις μη κυβερνητικέ οργανώσει από ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν. Αλλά οι γυναίκες ε, συνεχίζουν να αποτελούν την πλειοψηφία στον κόσμο των ε, ατόμων που υποφέρουν από την πείνα και την ένδια. Ε, και τελειώνει το παράθεμα. Τώρα οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται και σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε ευρωπαϊκό. Συμβαίνει εξάλλου αυτό και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπήρξε αύξηση της συμμετοχής των γυναικών αλλά πάν, βρισκόμαστε κάτω από το 35%. Οι γυναίκες ε, είναι πολύ πιο πολυάριθμες, π.χ. στα πανεπιστήμια από ότι άντρες, αλλά δύσκολα μπορούν να ανέλθουν στα ανώτατα επίπεδα της ακαδημαϊκής σταδιοδρομίας. Υπάρχουν πάρα πολλά τυχεία στο τομέα της ιατρικής ε, ή και σε άλλους κλάδους, αλλά σπάνια ανεβαίνουν την, ε, η αρχική κλίμακα. Υπάρχει λοιπόν πάντα κάτι το οποίο εμποδίζει τις γυναίκες στην ε, βελτίωση της τα γυναικών και ανδρών θα πρέπει να το, να το είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να δούμε και από μια διαφορετική άποψη. Μια γυναίκα αναφίβολα υφίσταται διακρίσεις ε, σε σχέση με τους άνδρες. Μια γυναίκα ε, έγχρωμη είναι, ε, υφίσταται μάλλον διακρίσεις σε σχέση με έναν ε, άντρα έγχρωμο. Και βλέπουμε στις διάφορες ανακοινώσεις, τα μέσα ενημέρωσης κλπ. Όλα αυτά τα στοιχεία. Βλέπουμε επίσης ποιο τρόπο χρησιμοποιείται η γυναίκα από τον τύπο και ειδικά από διαφημίσεις. Αυτές λοιπόν οι διακριτικές μεταχειρήσεις τις οποίες υφίστανται οι γυναίκες και τις οποίες διαπιστώνουμε λίγο πολύ παντού, αυτές οι μορφές λοιπόν ε, διακριτικής μεταχείρισης ε, το είναι κάτι το οποίο βλέπουμε και στο ζήτημα της ε, κοινωνικής ενημέρωσης και αυτό με τη σειρά του δημιουργεί μια άλλη μορφή διάκρισης το πώς οι υποψήφιες γυναίκες ε, αντιμετωπίζονται από τους ε, υποψηφίους, ε, από τους πολίτες, από τους εκλογείς. Οι γυναίκες έχουν λιγότερη προβολή σε σχέση με τους άνδρες και τα πλεονεκτήματα τα οποία έχει μια υποψηφιότητα γυναίκας δεν προωθούνται αρκετά. Οι γυναίκες υποψηφίες δεν αξιολογούνται για τις ικανότητές τους, για τις δραστηριότητες κλπ. Αν είναι λίγο πολύ ικανές να ασκήσουν τα καθήκοντα του βουλευτή. Στις περισσότερες περιπτώσεις ο τύπος ασχολείται με την προσωπική ζωή, με την οικογενειακή ζωή, με την ε, παρουσία τους, με το ενκόμωσή τους, με το φαίνεστε λοιπόν και όχι με το είστε ενώ οι άνδρες ε, προβάλλονται πάνω σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια, την οικονομία κλπ. Ε, οι γυναίκες ε, θεωρούνται ότι είναι πολύ πιο ευαίσθητες για αισθήματα που άπτονται της υγείας, του πολιτισμού κλπ και έτσι οι πολίτες πείθονται ότι οι γυναίκες δεν είναι εξίσου προετοιμασμένες όπως οι άνδρες για να κυβερνήσουν και την κατάλληλη στιγμή λοιπόν της επιλογής ο ε, εκλογέας ε, ψηφίζει άνδρα. Και θα σας αναφέρω μια περίπτωση που ίσως να γνωρίζετε. Όταν η Μισελ Μπασλέ εξελέγει πρόεδρος της Χιλής, μία από τις πρώτες ερωτήσεις που οι δημοσιογράφοι της έκαναν ήταν η παρακάτω. Τώρα εσείς πώς θα μπορέσετε να συμβιβάσετε και να συνδυάσετε τα καθήκοντά σας με τις οικογενειακές σας υποχρεώσεις, μητέρα, συζύγου κλπ. Κοιτάξτε, αυτό το ερώτημα δεν ε, έγινε ποτέ, δεν επιφύθηκε ποτέ σε έναν άνδρα πρόεδρο. Τον Μπαράκ Ομπάμα κανείς δεν τον ρώτησε πώς ε, προτίθεται να συνδυάσει τα καθήκοντά του ως Προέδρου με τα καθήκοντα του πατέρα δύο κοριτσιών και συζύγου και να σας αναφέρω τώρα και την προσωπική μου εμπειρία. Εγώ υπήρξα πρόεδρος της, στην Σύντρα το εμπορικό επιμελητηρίο. Είναι, το δεύτερος, είναι ο δεύτερος σε μέγεθος δήμος της Πορτογαλίας. Τα μέλη λοιπόν αυτού του Δημοτικού Συμβουλίου, του ε, ε, είναι σχεδόν όλοι άντρες και μετά από την εκλογή μου ως Δημοτική Συμβούλου και που επανειλημμένα μου ρωτήθηκα πώς αισθάνεστε εσείς επικεφαλής ενός Δημοτικού Συμβουλίου που αποτελείται από άνδρες αλλά μια τέτοια ερώτηση ποτέ δεν την κάνει κανείς σε άνδρα. Οι δημοσιογράφοι, τα μέσα ενημέρωσης θεωρούν ότι ο άνδρας διατάσσει και η γυναίκα υπακούει. Αλλά όταν τα πράγματα αλλάζουν και οι γυναίκες διοικούν και ε, δίνουν τις εντολές τότε ε, δίνονται αυτές, ε, γίνονται αυτές οι ερωτήσεις. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, πρέπει να καταπονημήσουμε αυτά τα στερεότυπα. Η γυναίκα μπορεί είναι χρήσιμη για να δουλεύει, αλλά όχι για να κυβερνά και να αποφασίζει. Νομίζω ότι αυτό είναι μια απέτηση της δημοκρατίας. Οι ποσοστά μας δείχνουν ότι η αύξηση των ποσοστών οδήγησε σε μια πιο δημοκρατική και πιο αρμονική κοινωνία. Ε, θα πρέπει λοιπόν να υπάρξουν νόμοι, την ισότητα των φίλων. Υπάρχουν φυσικά τέτοιοι νόμοι τόσο στην Πορτογαλία όσο και στην Ισπανία. Άνδρες και γυναίκες είναι απαραίτητες στην ε, δημόσια ζωή αλλά και στην ειδική φυσικά και όλοι έχουν τις υποχρεώσεις τους και τα καθήκοντά τους και τα δικαιώματά τους. Εδώ δεν πρόκειται για ένα πόλεμο φίλων, είναι ένας αγώνας ο οποίος θα πρέπει να ε, προχωρήσει παράλληλα προωθούμε τόσο από τους άνδρες όσο και από τις γυναίκες. Ευχαριστώ και τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Σούζαν Μπαντούτσι που θα μας κάνει μια παρουσίαση σχετικά με την εξαίρεση μιας κλασικής περίπτωσης αυτής των αποτελεσμάτων μιας μελέτης σχετικά με τη συμπεριφορά των μέσων ενημέρωσης ενάντια των γυναικών υποψηφίων. Ε, η κυρία Μπαλντούτσου έχει το λόγο. While the slides are ενώ ετοιμάζεται το μηχάνημα θα ήθελα να σας πω ότι ονομάζομαι Σούζαν Μπαλντούτσι και θα ήθελα να ευχαριστώ και τον Μαρελογίστα που με βοήθησε για αυτή τη σημερινή παρουσίαση και ετοίμασε τις ε, διαφάνειες για τη σημερινή παρουσίαση. As was uh, mentioned, talk to you about today. Όσο ελέγχθη, ο ρόλος των γυναικών σαν πολιτική υποψήφοι και ιδίως όσον αφορά την κάλυψη των νέων μέχρι τις ευρωεκλογές του 2009. Η έρευνα που έχω κάνει ε, οφείλεται εις, ε, τη, εις την κοινή γνώμη και τις δημοσκοπήσεις που παρουσιάστηκαν στις προηγούμενες ε, ομιλίες διότι εάν δείτε το, τους μέσους όρους βλέπουμε ότι υπάρχει λιγότερο πολιτικό ενδιαφέρον λιγότερη εμπλοκή με την Ευρωπαϊκή Ένωση άρα τι εξηγεί αυτές ε, τις διαφορές οι οποίες υπάρχουν ε, ε, έχει κάποια σχέση με τον οποίο προβάλλεται το θεσμικό όργανο, δηλαδή με την εκπροσώπηση των γυναικών στο θεσμικό όργανο και εάν το θεσμικό αυτό όγραφο ε, θεωρηθεί πιο θελκτικό για τις γυναίκες θα υπάρξουν περισσότερες ε, ενδιαφερόμενες για την πολιτική, για τις πολιτικές που προέρχονται από αυτό το θεσμικό όργανο. Αλλά επαρκεί διότι το θέμα δεν έχουμε 40-50% γυναικών που θα συμμετέχουν αλλά τι ε, καταλήγει από αυτή την εκπροσώπηση στους στους πολίτες και στα μέσα ενημέρωσης. Δηλαδή η, τα μέσα θα πρέπει να παρουσιάσουν τις γυναίκες, να δείξουν τι κάνουν οι γυναίκες για την εκπροσώπηση των γυναικών και για την εμπλοκή των γυναικών στην πολιτική και γι' αυτό το λόγο καταρτήσαμε αυτή την παρουσίαση και ο στόχος μου εδώ είναι να περιγράψω πώς προβάλλονταν οι γυναίκες το 2009 στις ε, ευρωεκλογές ποιες ήταν οι θέσεις τους ε, στους εκλογικούς καταλόγους, πόσες ε, υπήρχαν στις λίστες και να δούμε την ε, επίπτωση της εκπροσώπησης ε, ε, προς το γυναικείο φύλλο γενικώ. Σαν λοιπόν ε, υποψήφιες ευρωβουλευτίνες αυτό το οποίο ξέρουμε για την ε, προεκλογική εκστρατεία του 2009 σε όλα τα κράτη-μέλη, σε 27 κράτη-μέλη ε, εξετάσαμε πολλές ιστορίες και από όλες τις χώρες περίπου 35% των υποψηφίων ήταν γυναίκες και ε, ήταν 34% ε, από τους ε, υποψήφιους οι οποίες εξελέγησαν και 35% ε, εξελίξαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά άλλες ε, οι υποψήφιες οι οποίοι, ε, από τους άλλους υποψηφίους όπου υπήρχαν στις, ε, στα μέσα ενημέρωσης και δεν εξελέγησαν, μόνο 19% ήταν οι γυναίκες. Δηλαδή δεν ήταν ψηλά στο κατάλογο, ε, υπήρχε λιγότερο ποσοστό εκλογής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το πιο βασικό ήταν ότι δεν προβάλλονταν αρκετά στην ε, ενημέρωση του κοινού μετά τις εκλογές. Ποιες είναι οι επιπτώσεις αυτής της περιορισμένης ορατότητος. Όπως ξέρετε τα μέσα ενημέρωσης είναι σημαντικά για την ε, πληροφόρηση των πολιτών, συνδέουν τους πολίτες με τα θεσμικά όργανα και υπάρχει κάλυψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είναι σημαντική όπου λέγεται ποιος έχει δύναμη στο θεσμικό ε, όργανο και τι θέλει να κάνει. Εάν λοιπόν ε, το θεσμικό ε, όργανο δεν ασχολείται με τους πολίτες που εκπροσωπεί μπορεί να υπάρξουν επιπτώσεις και αυτό να έχει σχέση και με τη θέση των γυναικών. σε αυτή την διαφάνεια βλέπουμε τις γυναίκες εκπροσώπους και η γαλάζια γραμμή ε, ε, αναφέρεται στις γυναίκες οι οποίες είναι ε, στο ανώτερο τρίτο των υποψηφίων και εδώ αναφερόμαστε σε όλες τις πολιτικές ομάδες. Δεν φτάνει δηλαδή μια πολιτική ομάδα να περιέχει υποψήφιες γυναίκες αλλά να τις έχει και σε καλές θέσεις και βλέπετε ότι στις περισσότερες ε, χώρες ε, όσον αφορά τις ε, γυναίκες δεν κοιτάμε μόνο αν περιλαμβάνονται αλλά και τη θέση τους στον κατάλογο και στις περισσότερες χώρες που ήταν ήδη κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως πριν το 2004 οι γυναίκες είναι σε χαμηλές θέσεις εκτός από τη Δανία και στην Ελλάδα και υπάρχουν ε, σε αυτές τις δύο χώρες ε, οι γυναίκες που είναι πιο καλά τοποθετημένες. Στην Ιταλία παραδείγματος χάρη 36% ήταν γυναίκες αλλά μόνο 21% ήταν στο ανώτερο τρίτο. Στην Πορτογαλία μία παρεμφερής εικόνα. εις ε, ε, της ε, στην μετά το, στις χώρες οι οποίες έγιναν μέλη μετά το 2004 βλέπουμε λιγότερα, λιγότερες γυναίκες υποψήφιες και βλέπουμε ότι ήταν και μικρό το ποσοστό της συμμετοχής και μικρό το συμμετοχή το ποσοστό των γυναικών που ε, τις τοποθετεί στο ανώτερο τρίτο του καταλόγου. Αλλά όπως ελέγχθη προηγουμένως, οι γυναίκες δεν προβάλλονται, είναι χαμηλά στον κατάλογο και έχουν λίγες πιθανότητες να εκλεγούν. Θα ήθελα τώρα να αναφερθώ εις ε, την προβολή των ε, γυναικών υποψηφίων στα νέα και να σας περιγράψω πώς προβήκαμε στις μετρήσεις. Ε, είδαμε δηλαδή 60.000 ιστορίες τις τρεις τελευταίες εβδομάδες πριν τις εκλογές. Είδαμε ποιοι είχαν περιληφθεί, αν ήταν υποψήφοι για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να δούμε πόσες υποψήφοι εμφανίστηκαν εις ε, τις ευρωεκλογές και να αξιολογήσουμε για να δούμε αν τελικά οι γυναίκες εκπροσωπούνται ε, δίκαια στο ποσοστό μέχρι τις εκλογές. Είδαμε λοιπόν ότι το ποσοστό ήταν μικρό και δεν, υπήρχε μεγάλη προβολή των γυναικών στα μέσα ενημέρωσης. Αλλά στη Σουηδία αντιθέτως 50% των γυναικών ήταν στο ανώτερο τρίτο του καταλόγου ε, και υπήρχε ένα σημαντικό ποσοστό. Στην Ιρλανδία και στη Ρουμανία υπήρχαν περισσότερες γυναίκες ε, πάνω από το 1 τρίτον και αυτό οφείλεται σε δύο γυναίκες πολιτικούς οι οποίοι ήταν η μία ε, επικεφαλής ε, του καταλόγου και στη Ρουμανία επίσης βλέπουμε να υπάρχει ε, σημαντική προβολή. Σε άλλες χώρες όμως ε, υπήρχε πολύ χαμηλότερη προβολή και οι γυναίκες δεν ξεπερνούσαν το 20%. Η προβολή έχει σχέση με την θέση των γυναικών στον κατάλογο για να δούμε ε, αν θα υπάρχουν περισσότερες υποψήφοι, περισσότερες υποψήφοι στα νέα, στην ε, ε, ενημέρωση και ε, βλέπουμε ότι στην Ισπανία 4% μόνο των γυναικών εμφανίζονται στην τηλεόραση ενώ 42% των υποψηφίων ήταν γυναίκες. Ε, το Ηνωμένο Βασίλειο 19 των υποψηφίων ήταν γυναίκες αλλά μόνο 8% ε, παρουσιάζοντουσαν στις τηλεοπτικές εκπομπές Γενικώ λοιπόν θα περιμέναμε να υπάρχουν περισσότερες γυναίκες οι οποίες να προβάλλονται και περισσότερο στα νέα. Προτού τώρα μιλήσουμε για τις επιπτώσεις, θα ήθελα να αναφερθώ σε ορισμένους παράγοντες και να αναφερθώ στη σημαντική επίπτωση που μπορεί να έχει αυτό το γεγονός διότι οι γυναίκες μπορεί να είναι υποψήφιες αλλά δεν, είναι, δεν προβάλλονται στα νέα τι επιπτώσει έχει αυτό να δούμε δηλαδή εάν υπάρχουν άνθρωποι που αισθάνονται ε, υπεύθυνοι για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εάν ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπολογίζει τη γνώμη τους διότι ε, πολλές γυναίκες θεωρούν ότι πρέπει να εισακούονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενώ ε, 33% των ανδρών διαφωνούν. Μπορείτε να συγκρίνετε αυτή τη στατιστική με την στατιστική που παρουσίασα προηγουμένως όπου 39% των γυναικών θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπεύθυνη. Βλέπουμε λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πιο υπεύθυνο από ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπάρχουν περισσότερες γυναίκες ε, από ότι υπάρχουν ε, στο ε, από ότι υπάρχουν γενικότερα. Θα ήθελα λοιπόν εδώ να αναφερθώ εις την προβολή των γυναικών στα νέα και να σας πω ότι τα στοιχεία που αναφέρω ε, προέρχονται από μία μελέτη η οποία έγινε από το Ευρωβαρόμετρο μετά τις εκλογές. Εάν λοιπόν η προβολή είναι σημαντική, πώς μπορούμε ε, να έχουμε περισσότερες εκπροσώπους στις πολιτικές ομάδες, να είναι ψηλά στην, στον κατάλογο των υποψηφίων. Πρέπει όμως να δούμε πώς υποκινούνται και οι υποψήφιες ε, για να ε, ενδιαφερθούν για τις εκλογές και στα, αφού είδαμε την κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης εξετάσαμε και τους ευρωβουλευτές και τους ρωτήσαμε ε, ποιος τους προέτρινε να υποβάλουν υποψηφιότητα για την Ευρωβουλή και είδαμε εκεί τις διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών ως προς το πώς απάντησαν εις ε, την ερώτηση αυτή άλλοι είχαν πει είχαν κάνει ε, θετική απάντηση Βλέπουμε όμως ότι οι γυναίκες ε, είχαν ενθαρρυνθεί περισσότερο από περιφερειακά και τοπικά κόμματα. Η εθνική ομάδα, το εθνικό κόμμα, το, ο σύντροφός τους ή ο σύζυγος, άλλα μέλη της οικογενείας, η ομάδα ε, της κοινότητας, ε, ο ισχύων ευρωβουλευτής ενώ βλέπουμε ότι υπάρχουν διαφορές σε πολλά θέματα μεταξύ της θέσης μεταξύ γυναικών και ανδρών. Οι γυναίκες λένε ότι ενθαρρύνθηκαν από τον άντρα τους κατά 37% ενώ οι άντρες λένε ότι οι γυναίκες τους ενθάρρυναν μόνο κατά 23%. Υπάρχουν άλλες περιπτώσεις όπου φαίνεται κανείς δεν τους ενεθάρρυνε και ήταν απλούστατα μία προσωπική φιλοδοξία. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πώς οι γυναίκες και οι άντρες αντιμετωπίζουν διαφορετικά το θέμα το, της πολιτικής υποψηφιότητας ενώ οι γυναίκες οι άντρες θεωρούν ότι δεν χρειάζεται να τους εθαρρύνει κανείς για να προχωρήσουν και να προβληθούν. Καταλήγοντας, θα ήθελα να σας πω ότι νομίζω ότι είναι βασικό και να αυξήσουμε τον αριθμό των γυναικών υποψηφίων, να είναι σε καλύτερη θέση στους καταλόγους και να αυξήσουμε την προβολή τους ε, στα μέσα ενημέρωσης. Αυτό είναι βασικό για τα θεσμικά όργανα διότι οι γυναίκες αποτελούν το, από το 1 τέταρτο έως το ίμιση, 1 τρίτον ως το ίμιση των υποψηφίων ορισμένες ε, ε, είναι σε ε, δυσμενή θέση διότι είναι χαμηλότερα στον κατάλογο δεν έχουν τόση προβολή στα μέσα ενημέρωσης και τέλος τα πολιτικά κόμματα παίζουν μεγάλη σημασία στην πρόθεση των γυναικών σαν υποψηφίων. Foi uma apresentação muito interessante. Πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίασή σα. και επιβεβαιώνει τι ε, ανησυχίε μου και όχι μόνο καταδεικνύει εξάλλου και την προσωπική μου εμπειρία πάνω στο ζήτημα. Επίσης ε, πιστεύω πως θα μπορούσαμε καταλήγοντας να πούμε ότι υπάρχουν πολλά κράτη-μέλη τα οποία δεν υπάρχει ε, μια νομοθεσία που να παροτρύνει την ισότητα των φίλων. Εντάξει, οι λίστες ναι μεν περιέχουν πολλές γυναίκες αλλά στο τέλος ε, λίγες είναι αυτές που εκλέγονται. Και αυτό πολύ συχνά διότι οι γυναίκες αυτές ε, δεν μπαίνουν πάνω στην, ε, στη λίστα αλλά πολλές φορές στις τελευταίες θέσεις. Γι' αυτό λοιπόν και έχουν μεγάλη σημασία οι νόμοι περισσότητες διότι εκεί ορίζεται ποια θα πρέπει να είναι η θέση την οποία θα πρέπει να καταλαμβάνουν τα διάφορα φύλλα σε μια λίστα. Π.χ. θα μπορούσαμε να πούμε ότι υποψήφιος ε, θα πρέπει ε, μάλλον στο λίστα θα πρέπει να εναλλάσσονται άνδρες γυναίκες έτσι βεστώσει να μπορούμε να εγγυόμεθα πλέον ένα 33 ε, έως και 50% κάθε ένα, ένας άνδρας μια γυναίκα ή κάθε δύο άνδρες μια γυναίκα ε, επίσης γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ε, και μάλλον σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις επικεφαλής των λίστας βρίσκεται άνδρας. Και να υπενθυμίσω εδώ μια δήλωση που είχε γίνει ότι και που μας προβληματίζει. Όλα είναι συνδεδεμένα μαζί τους, όλα συνδέονται και πώς είναι δύσκολο να διακόψουμε αυτόν τον φαύλο κύκλο, αν θέλετε, στον οποίο έχουμε καταλήξει. Διότι λέγεται πως ειναι δυσκολο να διακοψουμε αυτον τον φαυλο αν θελετε τον οποιο εχουμε καταληξει διοτι λεγεται πως οσο πιο διάσημη είναι μια γυναίκα, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχει φυσικά να μπει σε, ψηλές, σε ψηλή θέση στην λίστα. Αλλά για να είναι διάσημη, να είναι γνωστή και αναγνωρισμένη, αυτό απαιτεί τα, μέλη, τα μέσα ενημέρωσης ε, να τις δώσουν την απαραίτητη προβολή. Καταλαβαίνετε λοιπόν πως ε, όπως σας είπα βρισκόμαστε ενώπιον ενός φαύλου κύκλου από τον οποίο πολύ δύσκολα μπορεί να εξέλθει κανείς. Είναι μια δυναμική η οποία δύσκολα μπορεί να καμφθεί. Θα έλεγα να ξεκινήσουμε τη συζήτηση και να αρχίσω εγώ με μια ερώτηση. Υπάρχουν ε, μελέτες ε, σχετικά με την παρουσία των υποψηφίων γυναικών ε, στα κοινωνικά δίκτυα, στα blog, διότι τα πράγματα έχουν αλλάξει. Δεν είναι όπως ήταν. Οι μορφές επικοινωνίας έχουν αλλάξει άρδιν παρουσία των ε, υποψηφίων δεν θα πρέπει να περνάει μόνο μέσω από την τηλεόραση, το ραδιόφωνο και τον ε, έντυπο τύπο, αλλά καλό είναι να περνάει και μέσω των ε, blog. Γι' αυτό λοιπόν είναι ενδιαφέρον να γνωρίζουμε κατά πόσο υπάρχει παρουσία σημαντική των υποψηφίων γυναικών σε αυτά τα νέα μέσα επικοινωνίας, κάτι το οποίο επηρεάζει τις το εκλογικό σώμα. Εγώ δεν γνωρίζω, αλλά θα τολμούσα να πω πως υπάρχει αύξηση στον αριθμό των γυναικών σε αυτά τα κοινωνικά δίκτυα και πως η διάδοση διαφόρων μηνυμάτων που αφορούν στις εργασίες και στις δραστηριότητε των γυναικών αυτών φτάνει σε υψηλότερο αριθμό αναγνωστών και μπορώ να πω πως πρόκειται για ένα φαινόμενο πολύ σημαντικό διότι με αυτόν τον τρόπο οι γυναίκες δεν ε, υπόκεινται σε διακριτική μεταχείριση διότι μπορούν ε, να έρθουν άμεσα και απευθείας σε επαφή με ένα μεγάλο ποσοστό ε, εκλογικού σώματος και έτσι να συλλέξουν περισσότερες ψήφους. Σας ευχαριστούμε για την παρέμβασή σας. Ε, πραγματικά ε, ακούσαμε πολύ ενδιαφέρουσες ε, ιδέες. Ε, η μελέτη αυτή θα μας προβληματίσει. Αν θέλετε να απαντήσετε στην ερώτησή μου, διαφορετικά να περάσουμε στη συζήτηση για να ακούσουμε αν και κατά πόσο υπάρχουν περαιτέρω ερωτήσεις. Δύο σκέψεις. Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για τα σχόλιά σας. Πρώτον, δεν είναι μια πολύ καλή ιδέα, αλλά εμείς τόσο συλλέξαμε τα στοιχεία από ε, υποψηφίους σχετικά με το ποια μέσα χρησιμοποίησαν στις, στην προεκλογική εκστρατεία. Έχουμε κάποια στοιχεία τα οποία δεν μπόρεσα ακόμα να αναλύσω. πολύ καλή ερώτησή σας και φυσικά θα ήταν ενδιαφέρον. Δεύτερον, είναι η σχέση μεταξύ αυτών των δραστηριοτήτων και των ε, δραστηριοτήτων των πολιτών. Ο τρόπος με τον οποίο ε, στρατεύονται οι πολίτες ε, σχετικά με πολιτικές διότητες αλλά και μορφές ενημέρωσης θα έλεγα γίνεται με τρόπο παθητικό. Δηλαδή, πολίτες δεν αναζητούν να ενημερωθούν αλλά παθητικά ενημερώνονται. Ο τρόπος επικοινωνίας με τους πολίτες ε, είναι ο Πρέπει να υπάρχει πολλή πληροφόρηση να ε, επιλέγεται από τα μέσα ενημέρωσης και οι πολίτες να μπορούν τυχαία θα έλεγα να πέσουν πάνω στην ενημέρωση. Με άλλα λόγια λοιπόν, αυτή η παθητική απορρόφηση πληροφόρησης ε, οφείλεται στη, ότι υπάρχει πάρα πολύ προφορία διαθέσιμη. Οι γυναίκες λοιπόν πρέπει να καταβάλουν προσπάθεια ώστε τα μηνύματά τους να περνάνε μέσω του τύπου και τηλεόρασεων. Είναι λοιπόν πολύ πιο δύσκολο για τους πολίτες να απορροφούν αυτές τις προφορίες παθητικά όσο λιγότερο οι προφορίες υπάρχουν. Και για τις γυναίκες είναι αυτές είναι λιγότερες. Ποιος επιθυμεί να λάβει το λόγο και να συμμετάσχει στη ζήτηση, Λίγα λεπτά μας απομένουν για την ολοκλήρωση αυτού του τμήματος. Δεν βλέπω να ζητάει κανείς το λόγο. Στο σημείο αυτό τότε θα μπορούσαμε να διακόψουμε για λίγο Κάνουμε λοιπόν μια διάλειμμα για καφέ και θα ξεκινήσουμε τις δραστηριότητές μας στις 4, σε ένα τέταρτο.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 Αγαπητοί φίλοι, μπορούμε να ξεκινήσουμε ή μάλλον να επαναλάβουμε τις εργασίες μας. Διαφέρουσες οι εισηγήσει και ο, και ο διάλογος που προξενήθηκε ε, και ερχόμαστε τώρα στο τρίτο τελευταίο μέρος και στην συμπερασματικό κομμάτι της σημερινής μας ημερίδας που έχει να κάνει με τα μέσα επικοινωνίας που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να ενισχύσουμε το διάλογό μας με τις γυναίκες και με τελικό στόχο να τις φέρουμε πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πάντα με την αμφίδρομη σχέση οι γυναίκες να έρθουν πιο κοντά στην Ένωση και η Ένωση πιο κοντά στις γυναίκες. Μόνο τότε μπορούμε να πούμε ότι γίνεται ουσιαστικός και αποδοτικός ε, το έργο μας. Ε, έχουμε την ε, ευκαιρία και το πλεονέκτημα να έχουμε μαζί μας <coughs> <coughs> I'm sorry. <coughs> να έχουμε μαζί μας εκπροσώπους από ειδικού οργανισμούς επικοινωνίας και είναι πραγματικά κάτι πολύ ενδιαφέρον για μας διότι συνήθως οι συνομιλητές μας είναι πολιτικοί από άλλους χώρους ή κοινωνική ε, κοινωνικοί εταίροι, ε, άνθρωποι που εργάζονται στη, ε, καθημερινά πώς να μεταδώσουν μηνύματα, να τα κάνουν αντιληπτά ή να καταλάβουν και οι ίδιοι τα μηνύματα της κοινωνίας και να τα αξιοποιήσουν. Δεν έχουμε πολύ, πολλές φορές αυτή την ευκαιρία και ευχαριστούμε τις παρεμβαίνουσες πολύ θερμά για αυτή τους την συμμετοχή σήμερα. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Βέρι Ντεβόσου,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 για την εισαγωγή. Νομίζω ότι είδατε ήδη πολλά νούμερα σήμερα. Δεν χρειάζεται να σας πω κι άλλα για τα νούμερα που ήδη ξέρετε. Θα προσπαθήσω να περάσουμε από τη θεωρία στην πράξη και θα προσπαθήσω να μιλήσουμε για ένα φαινόμενο το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τις γυναίκες σήμερα. Υπάρχει μια σοβαρή διαφορά μεταξύ των ε, μισθών των ε, ανδρών και των γυναικών. Αλλά θα ήθελα να σας πω ότι εγώ δουλεύω σε ένα γραφείο, σε μια ανεξάρτητη υπηρεσία, τη Mortier Brigade, εδώ στις Βρυξέλλες. Αλλά Η ουσία είναι ότι ειδικευόμαστε στο, στη σημασία για τον καταναλωτή. Σε αυτό ειδικευόμαστε και είναι κάτι το οποίο δεν άκουσα πολύ στην σημερινή συνεδρίαση. Θα εμβαθύνω λοιπόν σε αυτό. Είμαι λοιπόν ε, διευθύνων ε, σύμβουλος. Έχω ε, και συνεργάτες που είναι άντρες και συνεπώς ξέρω για τι πράγμα μιλάω. Θα σας μιλήσω λοιπόν για πέντε σημαντικούς κανόνες ε, επικοινωνίας, γιατί το να κάθεται κανείς απλώς και να μην λέει τίποτε δεν βοηθάει κανέναν. Ο πρώτος ε, κανόνας ε, που είναι πολύ σημαντικός είναι να πρέπει να βρει κανείς τι τον κάνει μοναδικό. Όταν μιλάμε για παράδειγμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τι το μοναδικό υπάρχει και ειδικότερα όταν μιλάμε για ένα θέμα όπως η μισθή. Και δεν θα πω σε πολλές λεπτομέρειες γιατί έχουμε ακόμη πολλά να κάνουμε. Ε, είναι όμως πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Θα ήθελα να σας μιλήσω λοιπόν για μια εκστρατεία. Είναι ένα οργανισμό για τον οποίο δουλεύουμε, το Equal Pay Day. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε αυτό το φαινόμενο, αλλά όταν ε, ένας άντρας ε, μετά από ένα χρόνο έχει ε, ένα συγκεκριμένο εισόδημα, η γυναίκα μετά για να έχει το ίδιο εισόδημα πρέπει να δουλέψει την ίδια χρονιά και ενδεχομένω παραπάνω. Και πρόκειται για μια ημερίδα που γίνεται το Μάρτιο ε, στις 26. Έχουμε λοιπόν πολύ χρόνο από τις 26 Μαρτίου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου για να δούμε τις εξελίξεις. Λοιπόν, μας ρώτησαν τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Αν μιλήσει κανείς ε, με τους άντρες και με τις γυναίκες ε, παραγνωρίζουν το πρόβλημα. Δηλαδή, εγώ ας πούμε δεν έχω κανένα πρόβλημα γιατί έχω τον ίδιο μισθό με τους ε, άντρες συναδέλφους αλλά αν δείτε πραγματικά τα χαρτιά υπάρχει σοβαρή διαφορά. Πρέπει λοιπόν να γνωστοποιήσετε καταρχά το πρόβλημα, να γίνει γνωστό ότι υπάρχει πρόβλημα όχι μόνο μεταξύ των γυναικών αλλά και στους άντρε. Επίσης πρέπει να ε, είναι γνωστό ότι έχει σημαντικό αντίκτυπο στην καθημερινή του ζωή. Θα μπω σε λεπτομέρειες ε, αργότερα και κάτι ακόμη και χαίρομαι πολύ που μιλάω για αυτό το θέμα σήμερα Πρέπει να γίνει κάτι οπωσδήποτε αν θέλουμε να υπάρξουν αλλαγές. Το πρώτο λοιπόν είναι τι σας κάνει μοναδικό και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το δεύτερο, μιλάμε πολύ για γεγονότα, θεωρία, νούμερα, αλλά άκουσα λίγα για τον καταναλωτή. Άκουσα κάτι, ότι, αλλά όχι αρκετά, γιατί πραγματικά αυτόν ενδιαφέρει πολύ αυτό το πρόβλημα. Πρέπει λοιπόν να δούμε ποια είναι η λύση στο πρόβλημά του. Και σε αυτό ακριβώς θα επισέλθω τώρα. τρία σημαντικά φαινόμενα έχω εντοπίσει. Το πρώτο είναι ότι οι διαφορές αρχίζουν από πολύ νωρίς. Γιατί ε, ένα αγοράκι παίρνει περισσότερο χαρτζιλίκι, για παράδειγμα, από ένα κοριτσάκι. Αυτό έδειξαν οι έρευνε. Για ποιο λόγο αρχίζει λοιπόν αυτό από την παιδική ηλικία. Υπάρχει λοιπόν μία εκστρατεία η οποία μας δείχνει ότι τα κοριτσάκια δεν έχουν καθόλου αυτοπεποίθηση. Tell me it's why the models look so perfect. Tell me I'm amazing, not because of how I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 όταν λοιπόν προσπαθήσετε, προσπαθήσετε να επικοινωνήσετε για πολύ συγκεκριμένα προβλήματα, πρέπει να γνωρίζετε τι συμβαίνει. Και το πρώτο σημαντικό γεγονός όταν μιλάμε για τις διαφορές είναι ότι αρχίζει, σε πολύ, ε, αρχίζει πολύ νωρίς αυτό. Οπότε μπορείτε να επικεντρώσετε την επικοινωνία σας ε, σε αυτό. Κάτι ακόμη. Οι τάσει των ρόλων. Θα σα πω μια ιστορία δεν ξέρω αν τη γνωρίζετε, ένας ε, πατέρας και ένας γιος, ε, ο πατέρας είναι στο τιμόνι και οδηγεί και γίνεται ένα ατύχημα. Πεθαίνει ο πατέρας, ο γιος μεταφέρεται στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, μπαίνει στο χειρουργείο, έρχεται ο χειρουργός, βλέπει το παιδί και λέει «Δεν μπορώ να τον χειρουργήσω, γιατί είναι ο γιος μου». Πώς είναι δυνατόν αυτό. Γνωρίζει κανείς. Ξέρετε, είναι επειδή είναι γυναίκα. Είναι η, είναι μητέρα. Εμείς πιστεύουμε ότι ο χειρουργός είναι οπωσδήποτε άντρας. Είναι λοιπόν ένα ψυχολογικό θέμα για το οποίο κάτι πρέπει να γίνει κάτι. Υπάρχει λοιπόν μια εκστρατεία που δείχνει ακριβώς ε, τα μοντέλα των ρόνων των ρόλων. Στο Βέλγιο, για την προσωρινή εργασία, και τοποθετεί τους άντρες ε, σε πολύ ελκυστική θέση. Ένα ακόμη βιντεάκι, το οποίο είναι πολύ πιο υπερβολικό. Ελπίζω να σας αρέσει. Ήθελα να σας το δείξω. Βλέπω ότι όλοι γελάτε. Μεταδόθηκε στο Βέλγιο και Τελικά μας είπαν ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε μετά από μία εβδομάδα στις ε, κάτω χώρες, ε, όμως ήταν αποδεκτό. Οι πολιτισμικές διαφορές λοιπόν είναι πολύ σημαντικό πράγμα όταν προσπαθεί κανείς να αλλάξει τα πράγματα. Επομένως το θέμα αυτό των ρόλων είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κάτι ακόμη είναι το θέμα του, του, είναι το γεγονός ε, που αφορά το δέσιμο των ε, ανδρών. Για παράδειγμα, πηγαίνω σε μια δεξίωση, υπάρχουν πάρα πολλοί άντρε και προσπαθεί κανεί ε, να δείξει κάποια κοινωνικότητα και είναι πάρα πολύ δύσκολο ε, και όλοι είναι ο ένα με τον άλλον και μιλάνε και έχει κανεί την εντύπωση ότι α, εγώ είμαι μια γυναίκα, ε, συγγνώμη που είμαι εδώ, αφήστε με να μπω στην ε, ε λέσχη σα την αποκλειστική. Είναι ενδεχομένω να, να πληρώνομαι λιγότερο, αλλά έχω τον ίδιο εγκέφαλο με εσά. Οπότε λοιπόν αυτό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 το οποίο ξεχνάμε συχνά είναι ότι πρέπει να ε, καταλαβαίνουμε την ομάδα στόχο και να επικοινωνούμε με τέτοιο τρόπο που τους κάνει να αισθάνονται ότι τους καταλαβαίνουμε. Ένας τρίτος κανόνας που είναι πολύ σημαντικός είναι το να είναι κανείς δημιουργικός γιατί πάρα πολλά ε, μέσα ενημέρωσης υπάρχουν. Ένας καταναλωτής λαμβάνει πάρα πολλά μηνύματα και δεν είναι εύκολο να τα αφομοιώσει όλα αυτά και αν, δεν υπάρχει δημιουργικότητα, ακόμη λιγότερο. Πρέπει να είμαστε δημιουργικοί για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε, να τραβήξουμε την προσοχή. Και είναι πολύ σημαντικό και ως προς τα τεχνικά μέσα που χρησιμοποιούμε. Θα ήθελα να σας δείξω τις εκστρατείες που κάναμε για το Equal Pay Day. Τέσσερα χρόνια δουλεύουμε για αυτούς. Και όταν ήρθαν πρώτη φορά σε εμά, ε, το πρώτο πράγμα που ήθελαν είναι η ευαισθητοποίηση, να γνωρίζει ο κόσμο ότι υπάρχει πρόβλημα. Το δεύτερο είναι η κινητοποίηση των γυναικών, να γνωρίζουν ότι υπάρχει μια διαφορά, ότι πρέπει να αντιδράσουν ε, για να γίνει κάτι. Και η εκστρατεία που θα αρχίσουμε σε μία εβδομάδα για τον διαφωτισμό των ανδρών. Δεν είναι μόνο δικό μας πρόβλημα, είναι και πρόβλημα των ανδρών, οπότε παρακαλώ κάντε κάτι. Το πρώτο θέμα λοιπόν, ευαισθητοποίηση. Το μήνυμα ήταν αν, είναι γυναίκα και πληρών, αν είστε γυναίκα και πληρώνεστε λιγότερο, είναι προσβολή. Δεν είναι μόνο προσβολή, είναι διάκριση. Οπότε παρακαλώ, αντιδράστε. Hey, bitch. Hey, John. Here's your report, Can. Thanks. Good morning. Hey.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 31 Μαρτίου ήταν η ημερομηνία αυτού του βίντεο. Το δεύτερο ήταν η εκστρατεία για να αντιδράσουν οι γυναίκες. Να γνωρίζει ο κόσμος και η κοινωνία ότι δεν είναι καλή η διαφορετική αμοιβή. Αν εγώ παίρνω 24% χαμηλότερο εισόδημα, αυτό σημαίνει ότι από τις 3 και 5 δουλεύω δωρεάν. Οπότε κάναμε ένα ραδιοφωνικό σποτάκι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 στις ε, γυναίκες ε, στις σελίδες ε, αναφερόταν ακριβώς ότι μετά τις 3 και 5 είναι σαν να δουλεύω δωρεάν και για τους άντρες ότι εγώ δεν θα δούλευα δωρεάν μετά τις 3 και 5. Όσον αφορά το διαφωτισμό των ανδρών. Μέχρι σήμερα νομίζω ότι όλος ο κόσμος παντού θεωρεί ότι είναι ένα πρόβλημα των γυναικών μόνο, αλλά δεν είναι αλλά δεν είναι γιατί οι άντρε ε, έχουν γυναίκες στη ζωή τους και αν δεν είναι η γυναίκα τους είναι η μητέρα του η κόρη του. Οπότε αν πληρώνετε λιγότερο αυτό έχει έναν αντίκτυπο στην καθημερινή σας ζωή των ανδρών. Οπότε αν θέλετε μια καλύτερη ζωή για εκείνες πρέπει να εξασφαλίσετε ότι υπάρχει ίση αμοιβή και για του άντρε και τι γυναίκε. Νομίζω ότι το μήνυμα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ότι όλοι επωφελούνται αν γίνει κάτι για την διαφορά των μισθών. Τέταρτος κανόνας και πολύ σημαντικός είναι να είναι κανείς συνεπής ε, όταν μιλάει για ένα πρόβλημα όταν είστε η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να μιλάτε με τέτοιο τρόπο που να δείχνετε ότι υπάρχουν συγκεκριμένες αξίες, ότι μπορεί να αλλάζει η διάθεση, αλλά εν πάση περιπτώσει το μήνυμα πρέπει να περνάει είναι ότι σας γνωρίζω, γνωρίζω το πρόβλημα και αν θέλετε να έχετε διαφορετική εκστρατεία από ό,τι τις προηγούμενες φορές πρέπει κάθε φορά να δείχνετε ότι προσεγγίζετε το πρόβλημα διαφορετικά. Όχι, δεν πρέπει να το κάνετε αυτό. Κάθε φορά που ε, θέλετε να επικοινωνήσετε, ε, προσπαθήστε να είστε σαφείς και συνεπείς, ε, με πνευματόδη, με έξυπνο τρόπο, αλλά να βλέπετε και την οπτική γωνία του καταναλωτή. Ξεκινήστε όχι βλέποντας τα πράγματα από τη δική σας πλευρά ως Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά από την πλευρά του καταναλωτή. Το κάνετε αυτό ήδη γιατί κάνετε κάποια έρευνα, αλλά προσπαθήστε να το κάνετε και στην πράξη. Κάτι ακόμη είναι ο διάλογο. Αν έχετε ένα ενδιαφέρον μήνυμα, θα το ακούσουν και θα προσπαθήσουν οι καταναλωτέ να μιλήσουν ε, μαζί σα και εκείνοι. Μην ε, είστε πάρα πολύ ε, διδακτική στην προσέγγιση σας. Ε, προσπαθήστε να είστε κάπως πιο πνευματώδεις, όχι όμως με πολύ παθητικό τρόπο να στέλνετε απλώς ένα μήνυμα και να ελπίζετε ότι ο κόσμος θα σας ακούσει. Προσπαθήστε να, προσπαθήστε να το κάνετε με ενεργητικό τρόπο, όχι με παθητικό. Και μην ε, μιλάτε ως... Ε, οργανισμός, προσπαθείτε να επικοινωνήσετε σαν άνθρωπος. Και ο πέμπτος κανόνας που είναι ο πιο σημαντικός ε, είναι γιατί κανείς προσπαθεί να είναι μοναδικός, δημιουργικός, ε, συνεπής και, και έχει μία σημασία. Γιατί θέλει να είναι αποτελεσματικός. Οι εκστρατείες Equal Pay Day από 25% είχαν ως αποτέλεσμα, είχε ως αποτέλεσμα να μειωθεί ο μισθός, η διαφορά του μισθού από 25% σε 23% είναι κάτι το οποίο έγινε γιατί ακριβώς γνώρισε επιπλέον, επιτέλους ο κόσμος το πρόβλημα. Ήταν γνωστό το πρόβλημα επιτέλους και χαίρομαι που σας το λέω σήμερα γιατί η πολιτική όντως μπορεί να οθήσει τα πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι λοιπόν σημαντικό να ευαισθητοποιηθούν όλοι και οι άνδρες κυρίως ότι είναι και δικό τους πρόβλημα. Εκεί λέει ότι οι γυναίκες όλο και περισσότερο πιο ψηλά να πρέπει να πηγαίνουν για να τις λαμβάνουν σοβαρά υπόψη. Εγώ φοράω πολύ ψηλά τα κούνια σήμερα για να φαίνομαι ψηλότερη. Ελπίζω ότι η κόρη μου δεν θα χρειάζεται να φοράει τα κούνια για να την παίρνουν σοβαρά υπόψη. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Ντεβός. Πραγματικά μας βγάλατε από το καθημερινό μας περίγραμμα και μας δώσατε την αφορμή να σκεφτούμε πράγματα, μεθόδους και πολλά εργαλεία που ίσως έχουμε αλλά δεν τα έχουμε αξιοποιήσει με, με, την κατεύθυνση της επικοινωνίας. Τώρα θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε ε, την κυρία ε, <clears throat> Ναταλή Τόντ, ειδική επίσης στην επικοινωνία, είναι από, τον, από την εταιρεία Ogilvy. Σας ευχαριστούμε πολύ. You have the floor. Λοιπόν, ώσπου να αλλάξουν οι διαφάνειες για τις παρουσιάσεις θα σας πω τι εργασία έχουμε κάνει σχετικά με την ε, επικοινωνία των πολιτών με τις ε, κοινοβουλευτικές ομάδες διότι είμαι υπεύθυνη στην Όγκυλβη για την επικοινωνία αλλά είναι μια εταιρεία η οποία ε, έχει σημαντική εμπλοκή στη διαφήμιση και γι' αυτό θα σας μιλήσω και για τα δύο θέματα η εργασία την οποία έχουμε κάνει από τις Βρυξέλλες είναι οι εκστρατείες ή να βοηθάμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει εκστρατείες για επαφή ε, με τις ε, γυναίκες, με τους πολίτες και πρέπει να ξέρουμε τι σας υποκινεί σαν καταναλωτή, σαν πολίτη ε, σε σχέση με ένα προϊόν και καταρχήν να κοιτάξουμε αυτά τα στοιχεία. Σήμερα άκουσα από ορισμένε ερωτήσεις και από άλλους ομιλητές ε, διάφορα θέματα τα οποία θα προσπαθήσω να ενσωματώσω στην παρουσίασή μου ε, ιδίως όσον αφορά το κοινωνικό πρόγραμμα και το πολιτικό πρόγραμμα την ανάγκη να επικοινωνούμε σωστά χρησιμοποιώντας τα σωστά μέσα και θα επανέλθω σε αυτό να η προσπάθεια προσπάθεια να καταρριφθούν ορισμένα στερεότυπα τα οποία υπάρχουν και ε, η προσπάθεια να δημιουργηθεί μία επαφή με τις γυναίκες σαν γυναίκες και όχι τόσο όσον αφορά την πολιτική χρειά τους. Θα αναφερθώ στο θέμα της διαφήμισης και ιδίως στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου έχουν γίνει μελέτες αυτές χωρίς όμως να υπερβάλλω ελπίζω. Καταρχήν λοιπόν πρέπει να δούμε ποιο είναι το κοινό μας ποιος είναι ο στόχος σας ε, και πώς μπορείτε να έρθετε σε επαφή με το στόχο αυτό πριν αρχίσετε να δραστηριοποιείτε. Να ξέρετε ποιο είναι το κοινό, το ακροατήριο και με ποιον τρόπο μπορείτε να κάνετε επαφή. Υπάρχουν ορισμένα θέματα τα οποία θα επιτρέψουν να έρθει κανείς σε επαφή με τις γυναίκες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να κοιτάξουμε και ποιες είναι οι προσδοκίες και τα ιδεώδη. Θα αναφέρω ορισμένα παραδείγματα. Καταρχήν όσον αφορά μία εκστρατεία για την υγεία ε, ε, και εστιασμό σε θέματα των καταναλωτών για να δούμε πώς αυτά σας προσεγγίζουν ή όχι. Καταρχήν λοιπόν θα ήθελα να σκεφτούμε ποιο είναι το κοινό στον οποίο αναφερόμαστε ότι οι γυναίκες είναι περίπλοκες, ζουν μια περίπλοκη ζωή είτε σαν μητέρες είτε σαν εργαζόμενες, σαν πολιτικοί, σαν κόρες. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε τι προσπαθούμε εμείς να μεταβιβάσουμε και πώς προσπαθούμε να το μεταβιβάσουμε και πρέπει να σκεφτούμε αυτές τις διάφορες ε, ε, ε, δυνατότητες επικοινωνίες τις οποίες χρησιμοποιούν οι γυναίκες δηλαδή που καταναλώνει την πληροφόρηση τα στοιχεία που είναι ο καλύτερος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να επικοινωνήσουμε και δεν είναι εξαντλητική η παρουσίαση αυτή απλούστατα να δούμε μέσω της τηλεόρασης των εφημερίδων των περιοδικών ε, ή άλλων μέσων ε, τα οποία πρόσκυνται στις γυναίκες. Αρχίζει το θέμα και περιπλέκεται όταν αρχίστε και σκέφτεστε τις ψηφιακές επικοινωνίες. Υπάρχουν όμως συγχρόνως και μεγαλύτερες δυνατότητες και η μία προηγούμενη επικεφαλής της συνεδριάσεως αναφέρθηκε σε αυτό διότι ε, εμείς ε, προσκύμεθα σε ορισμένους άλλους τύπους αλλά αυτό που διαπιστώνουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι ε, οι πιο δραστηριές είναι οι νέες μητέρες οι οποίες αισθάνονται ότι πρέπει να έχουν πιο στενές επικοινωνίες μέσω του διαδικτύου και προσπαθούμε να διοχετεύσουμε και από εκεί τις πληροφορίες μας και χωρισμένα στοιχεία εάν τα χρειαστείτε αργότερα. Για να πούμε και πάλι ότι μία γυναίκα είναι περίπλοκη και μέρος της κοινωνίας όταν ε, εξετάζουμε το θέμα ε, της ε, ισορροπίας μεταξύ εργασίας και ζωής πρέπει να δούμε τι εμφανίζεται στις διαφημίσεις, πώς παρουσιάζεται εκεί η γυναίκα συνολικά. Δηλαδή βλέπουμε ποια είναι η προσδοκία μας για την ισορροπία ζωής και εργασίας Προσπάθησα λοιπόν και πάλι να ε, ε, λύσω πληροφορίες από τους συναδέλφους ή στη διαφήμιση και να δούμε τι εμπνέει τη γυναίκα στη διαφήμιση. Πρόκειται για μία γυναίκα 32 χρονών, ξανθιά, η οποία περνάει σε ε, πολυσύχνα στους δρόμους φορώντας ένα κουστούμι, μυρίζοντας τριαντάφυλλα ξύλα κρατώντας ε, τσάντες ε, και ε, συγχρόνως είτε ανακατεύοντας το φαγητό ή δοκιμάζοντας φαγητό ή μιλώντας με φίλες της ή φορώντας μία μεταξωτή μπλούζα ίσως όλα αυτά σας φαρνούν στερεότυπα αλλά είναι στερεότυπα που χρησιμοποιούνται στη διαφήμιση και πρέπει να δούμε πώς θα απομακρυνθούμε από αυτά τα στερεότυπα και να ασχοληθούμε με ό,τι πραγματικά ενδιαφέρει τις γυναίκες, την πραγματικότητα δηλαδή ε, πώς, ποια είναι η πραγματικότητα και πώς αντιδρούν οι γυναίκες στην πραγματικότητα και θα σας δώσω μερικά βασικά στοιχεία. Είναι θέματα από την καθημερινή μας ζωή που μας αγγίζουν, που έχουμε μέσα μας και που επηρεάζουν την ανθρώπινή μας συμπεριφορά και τον τρόπο με τον οποίο ζούμε. Είναι θέματα τα οποία μας αγγίζουν στην καθημερινή μας ζωή θα κοιτάξουμε και τους διάφορους τύπους επικοινωνίας. Ξέρω ότι είναι αντιφατικό ε, να πούμε ότι οι γυναίκες είναι έτσι και οι άντρες είναι αλλιώς. Αλλά το θέμα κλειδί το οποίο με ενδιέφερε ήταν ε, ότι οι γυναίκες αμφισβητούν περισσότερο, ε, προσπαθούν να βρουν περισσότερα κοινά στοιχεία και να μοιράζονται, το οποίο είναι επίσης σημαντικό αν σκεφτείτε ότι και αυτός είναι ένας τρόπος να επικοινωνήσετε. Δηλαδή ότι το να μοιράζεσαι κάτι είναι ένας τρόπος επικοινωνίας. Και δημιουργικότητα για να επανέλθω στο θέμα αυτό. Οι γυναίκες είναι πολύ δημιουργικές στην καθημερινή του ζωή προσπαθούμε να βρούμε μία διασύνδεση, να βρούμε ένα νόημα και αυτό είναι θετικό, δεν είναι κακό. Γνωρίζοντας λοιπόν ότι οι γυναίκες συνεχώς προσπαθούν να σκέπτονται και να δρουν σε διαφορετικά επίπεδα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις διαπιστώσεις για να εμπλουτίσουμε την ε, ε, εξαρτία μας επικοινωνίας για να δημιουργήσουμε μια πιο στενή σχέση, να, κάνουμε, να δημιουργήσουμε μια επαφή. Προσπαθούμε λοιπόν να βρούμε τα πραγματικά προβλήματα τα οποία υπάρχουν και ε, είτε πρόκειται για την ισότητα της αμοιβή είτε για κάτι άλλο πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι το θέμα το οποίο προσπαθούμε να περάσουμε είναι βασικό και στη συνέχεια πρέπει να ερευνήσουμε ποια είναι η λύση και πώς θα μπορέσουμε να προσεγγίσουμε αυτή τη λύση μέσω των διαφόρων μεθόδων. Να προσπαθήσουμε δηλαδή δημιουργικά να προκαλέσουμε μία αλληλική συμπεριφοράς που είναι κάτι το οποίο βασίζεται εις το κοινωνικό μάρκετινγκ όπου η δημιουργικότητα μπορεί να επηρεάσει τα θέματα της συμπεριφοράς και μπορεί να επιφέρει αλλαγές. Τι κάνουμε στην εταιρεία μας τώρα στην Όγκυλβη. Κοιτάζουμε να βρούμε ποιες είναι οι φιλοδοξίες, οι προσδοκίες, να δούμε ποιες είναι οι προσδοκίες. Πού προσπαθείτε να καταλήξετε, ποιο είναι το μεγάλο ιδεώδες το οποίο έχετε. Πρέπει να, παλιά μιλούσαμε για μεγάλη ιδέα, big idea, τώρα μιλάμε για μεγάλο ιδεώδες, big ideal και αυτό αντικατοπτρίζει και το πρόβλημα μεν αλλά και μας δείχνει πώς θα πλησιάσουμε τη λύση. Θα σας δείξω λοιπόν πώς η εκστρατεία μας βασίστηκε στο στοιχείο αυτό και προχώρησε από, από εκεί. Παραδείγματος χάρη για μία κρέμα σώματος ε, μία διαφημιστική καμπάνια. Ε, μία ιδέα που είχαμε για τον Ντόβ είναι ότι πιστεύουμε ότι ο κόσμος θα είναι καλύτερος εάν και θα μπορούσαμε να πούμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιστεύει ότι ο κόσμος θα είναι καλύτερο εάν οι γυναίκες ήταν, δηλαδή ποιο είναι το αποτέλεσμα που επιδιώκεται. Επί του προκειμένου για τον ΤΟΒ, εάν οι γυναίκες αισθάνονται καλύτερα για τον εαυτό τους και αυτό βασίστηκε σε πάρα πολλή μελέτη η οποία εστιάζεται στην αυτοεκτίμηση των γυναικών. Αυτό είναι ένα θέμα που έφυγε και προηγουμένως και είχε εκπληκτικά αποτελέσματα διότι από τη μελέτη την οποία κάναμε στον Καναδά όπου ξεκινήσαμε ε, ένα μεγάλο ποσοστό των ε, ε, γυναικών θεωρούσαν ότι δεν είναι ούτε ωραίες ούτε θελκτικές και ήταν ανησυχητικό, τρομακτικό. Οι γυναίκες πρέπει να αισθάνονται καλά στο πετσί τους, να μπορούν δηλαδή να αισθάνονται ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία τις κάνουν ωραίες. Προσπαθώ λοιπόν να σας βοηθήσω να ακολουθήσετε την πνευματική μου διεργασία και γι' αυτό είπαμε ότι το πρώτο είναι να καταργήσουμε τα στερεότυπα. Ασχέτως ηλικίας, ασχέτως γενεάς, όπου και να βρίσκεστε, να αισθάνεστε ότι πρέπει να σας εκτιμούν, ότι πρέπει να σας θεωρούν ότι είσαστε ωραία και ε, έτσι αναπτύξαμε αυτή την εκστρατεία η οποία προσπάθησε να καταργήσει ορισμένα ταμπού, ορισμένες προκαθορισμένες ιδέες, να είναι κανείς ε, πιο ηλικιωμένος, να έχει φακίδες, να έχει διαφορετικό χρώμα δέρματος ε, προσπαθήσαμε λοιπόν να είμαστε πιο προκλητικοί και είχαμε, ε, ε, δημιουργήσαμε αμφιλεγόμενα αποτελέσματα διότι εις την Αμερική και ε, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ηνωμένο Βασίλειο μας είπαν οι υπεύθυνοι της ε, διαφημιστικής καμπάνιας ότι δεν θα ακολουθήσουμε αυτή την οδό και στο τέλος το δεχτήκανε ε, δηλαδή κάποιος είχε το σθένος να δημιουργήσει κάτι το οποίο θα προκαλούσε και θα κατέλειε τα στερεότυπα και αυτό έγινε σε πολλές χώρες τώρα διότι άπαξ και ε, μπόρεσε να επιτύχει σε δύο αγορές κλειδιά μπορέσαμε να το προωθήσουμε και αλλού όχι πάντοτε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο δεν μπορείτε να βάζετε παντού σε όλες τις χώρες τις ίδιες αφήσει, αλλά παίρνετε μία ιδέα της ποικιλία και των προκλήσεων οι οποίες ε, υπάρχουν. Οι διάφορες λοιπόν γυναίκες σε διάφορα μεγέθη, σε διάφορες ηλικίε είναι ένα θέμα το οποίο μας βοηθά να ξεκινήσουμε μία συζήτηση, να κρατήσουμε ανοιχτό το διάλογο και να αφήσουμε τις γυναίκες να αναθεωρήσουν τις θέσεις τους στο πλαίσιο αυτό. Να συμμετέχουμε λοιπόν σε συζητήσεις ακόμη και στο διαδίκτυο διότι ε, δεκάδες χιλιάδες γυναικών ασχολούνται με ε, την ε, ομορφιά και τι σκέφτονται και πάντη και πάλι εάν ασχοληθούμε στο διαδίκτυο υπάρχει δυνατότητα να ανταλλάξουμε blog και τα λοιπά βλέπετε ότι εδώ πρόκειται για μια πιο ηλικιωμένη ε, κυρία η οποία πάλι προσελκύει την προσοχή θέλω να σας δείξω επίσης τι έγινε για ε, ένα workshop που κάναμε για μητέρες και κόρες ε, και το χρησιμοποιήσαμε όχι όχι σαν διαφήμιση αλλά για το workshop αυτό για να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τις γυναίκες αυτές και τα παιδιά τους, τις κόρες τους να αυξήσουν την αυτοεκτήμασή τους και ε, υπήρξαν ε, ε, μηνύματα τα οποία βάλαμε σε διάφορους σταθμούς περιφερειακούς, τηλεοπτικούς και θα δείτε ένα βίντεο και πώς λειτουργεί όχι μόνο στο Good Morning America στην Αμερική αλλά και σε άλλα προγράμματα παρακαλώ λίγη υπομονή μέχρι ότου να ξεκινήσει το βίντεο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 Λοιπόν, για να σας δώσω μία ιδέα του τι κάνουμε. Και αυτό ήταν το ουσιαστικό βίντεο του 1997. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν είναι πάντοτε εύκολο να προβλέψετε τι θα γίνει με ένα βίντεο διότι δεν ξέρετε ποιον θα αγγίξετε. Ε, εάν λοιπόν πείτε θα κάνω ένα βίντεο για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να έχει αντίκτυπο, μπορεί και όχι. Εξαρτάται αν είσαστε ε, αστείοι, αν σοκάρετε ή ε, τι γίνεται. Ήθελα λοιπόν να σας δείξω αυτό διότι μιλάει για την ομορφιά αλλά συγχρόνως ασχολείται και ε, με τις διάφορες γενιές διότι το επόμενο βίντεο ασχολείται περισσότερο με τις νέες δηλαδή με τις μητέρες και πώς οι μητέρες αντιμετωπίζουν τα νέα κορίτσια και πώς αισθάνονται. Ελπίζω λοιπόν ότι θα σας ενδιαφέρει. Λοιπόν, ε, τώρα θα ασχοληθούμε με κάτι άλλο. Θα ήθελα δει στον υπόλοιπο χρόνο να ασχοληθώ με κάτι το οποίο ίσως σας ενδιαφέρει πιο πολύ, δηλαδή την Ευρωπαϊκή ε, Οργάνωση για την καταπολέμηση του καρκίνου. Ήταν ε, μία ε, εταιρεία η οποία προσπάθησε και νομίζω επιτυχώς να συνεργαστεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να επηρεάσει και να πλησιάσει τις γυναίκες. Εάν έχουμε χρόνο θα ήθελα να, να ασχοληθώ με αυτό. Πόσο χρόνο έχω ακόμη πόσο χρόνο μπορείτε να μου διαθέσετε. Yeah, okay, so we won't have time. <laughs> okay. Ωραία. Λοιπόν, το βασικό μήνυμα εδώ είναι ότι ο στόχος ήταν και ε, να ε, ενημερώσουμε τις γυναίκες και να τους δώσουμε τις δυνατότητες. Δηλαδή ε, να τις βοηθήσουμε να ενταχθούν σε προγράμματα προλήψεως και καταπολέμησης του καρκίνου του τραχύλου και να έχουμε μια επικοινωνία στα κράτη-μέλη και συγχρόνως να εμπλακεί και να συμμετάσχει και το ιατρικό επάγγελμα και αυτό έχει γίνει πριν από τέσσερα χρόνια ε, με μια ομάδα που ήταν, κατά της, που ήταν υπέρ της καταπολέμησης του καρκίνου. Ξεκινήσαμε λοιπόν εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ε, αναφέρθηκε στα μέσα ενημέρωσης και ε, ε, κάθε μέλος της οργάνωσης αυτής αισθάνθηκε ότι υπήρχε μία πολιτική όθηση και κίνηση την οποία μπορούσαν ε, να χρησιμοποιήσουν για την αγωγή, για την πρόληψη και την επόμενη η χρονιά ε, ασχοληθήκαμε μέσω του διαδικτύου στο facebook ε, με ε, διάφορες, διάφορα έγγραφα μπορούσε κανείς να κατεβάσει από το διαδίκτυο και ήθελα να σας δείξω ένα παράδειγμα τώρα το οποίο ίσως δεν είναι τόσο παραγωγικό αλλά το οποίο επέτρεψε στις γυναίκες αυτές να πιστεύουν ότι έχουν κάποιο ρόλο και κάνουν σωστή δουλειά δουλειά. Ε, αντιλαμβάνομαι βέβαια ότι κι εσείς θέλετε να βλέπετε αποτελέσματα σε αυτά που κάνετε. Ε, Όσον αφορά τις Ηνωμένε Πολιτείε, είχαμε ασχοληθεί για την καρδιοπάθεια στις γυναίκες χρησιμοποιώντας άλλες τεχνικές ε, χωρίς ε, τα μέσα ενημέρωσης αλλά με ε, role models και χρησιμοποιώντας και τη μόδα. Η μόδα όλο και περισσότερο ασχολείται με τέτοια θέματα πέραν των πολιτικών. Ε, και σε συνεργασία με εταιρείες τροφίμων εδώ, με τον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος, ε, ε, το οποίο σημαίνει ότι δεν είναι υποχρεωτικά θέματα δημοσίου συμφέροντος αλλά ε, μπορεί να συνεργαστούμε και με ιδιαιώτες και οι μέθοδοι αυτής αποδίδουν στις διάφορες χώρες πρέπει να είναι προσαρμοσμένες αλλά πρέπει να είσαστε ε, βέβαιοι ότι έχετε αντιληφθεί ποιο είναι το κοινό σας έχετε κάνει σωστά την έρευνά σας έχετε μια σωστή στρατηγική ε, και ε, ξέρετε πού θα μπορέσετε να κινηθείτε καλύτερα κατά τρόπον ώστε να χρησιμοποιήσετε καινοτόμες συνεργασίες, ε, δημιουργικά υλικά και εργαλεία και μία αξιολόγηση. Βεβαίως η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων είναι βασική. Ε, εδώ θα σταματήσω. Δεν ξέρω τι άλλο θα θέλατε, αλλά εγώ σας ευχαριστώ. Thank you very much for your presentation. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση. Αυτά που ακούσαμε και πραγματικά ξεφεύγουν από το περιεχόμενο των ε, σεμιναρίων και των συζητήσεων που έχουμε συνήθως. Μας δώσατε ε, και η, η κυρία Ντεβός και η κυρία Τόντ μας έδωσαν έναυσμα για προβληματισμό και για συζήτηση. Ο λόγος τώρα είναι σε εσά. Ποιος θέλει να απευθύνει μια ερώτηση. Ε, σας παρακαλώ λέγετε το όνομά σας και την ιδιότητά σας όταν παίρνετε το λόγο. Εσείς. You have the floor. Oui, bonjour. Marie Καλή σας ημέρα. Μαρή γραμμό. Είμαι βοηθός ε, του Μάρκου Τάραμπέλα. Ε, η παρουσίασή σας ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Θεώρησα πως πρόκειται για μια προσέγγιση εντελώς διαφορετική, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα σίγουρα, αλλά ασχολείται με πώς τα ευρωπαϊκά όργανα μπορούν να επικοινωνήσουμε το προς τα έξω. Αλλά το πρόβλημα ως βοηθού αλλά και του βουλευτή μου είναι να περάσουμε προς τα έξω τα, τι κάνουν οι ευρωβουλευτές για τις γυναίκες μέσω των μέσων ενημέρωσης. Όταν ξεκινήσαμε προσπάθησαν να έρθουν σε επαφή με τα γυναικεία περιοδικά, όλους τους ε, ε, δημοσιογράφους γαλλόφωνων εντύπων και πολύ λίγα άτομα βρήκα να ενδιαφέρονται, να ε, εξετάζουν το ζήτημα αυτό, ιδιαίτερα ό,τι τα γυναικεία πρεδικά. Ελάχιστο ενδιαφέρον. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να δεχτούμε τα διάφορε συμβουλέ σα, δημιουργική κλπ. Πώ μπορούμε να το κάνουμε, διότι οι βουλευτέ δεν μπορούν να ξεκινήσουν κάποιε εκστρατείε μεγάλη εμβέλεια όπω μπορείτε να το κάνετε εσεί. Τι μπορούν να κάνουν οι βουλευτέ λοιπόν για να προκαλέσουν το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωση αναφορικά με δικαιώματα των γυναικών και ισότητα των φύλων. Έχετε κάποια ιδέα και είμαι σίγουρη ότι <laughs> ήδη ε, απαντάει σε προβληματισμούς που έχουν και άλλοι βουλευτές και άλλοι ε, πολιτικοί παράγοντες σε εθνικό ή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Άλλη ερώτηση για να μπορέσουν να απαντήσουν ε, συλλογικά οι προσκεκλημένες μας από τις εταιρείε επικοινωνίας. Άλλη ερώτηση. Η κυρία Μωρά. Η Ευρωβουλευτής η κυρία Μωρά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ακούσαμε ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις εκτός ε, κοινού. Θα έλεγα εξής, ε, τι προβλέπετε για να μπορέσουμε να προωθήσουμε κάποιο πολιτικά μηνύματα σε 27 κράτη-μέλη. Είδαμε ότι υπάρχουν πολιτιστικές διαφορές και πως εσείς ε, στο επάγγελμά σας ε, αντιμετωπίζετε αυτές τις πολιτικές διαφορές χρησιμοποιώντα διαφορετικά μέσα σε συνάρτηση με την κάθε χώρα. Ε... Εμείς όμως ε, μπορούμε να στείλουμε ένα ενιαίο μήνυμα προς τα 27 κράτη-μέλη ε, δεν βρισκόμαστε ακόμα σε αυτό το στάδιο της ε, ταυτόσιμης ε, και μονοσήμαντης ενημέρωσης προς τα 27 κράτη. Κυρία Μωρά, ευχαριστούμε πολύ για την ερώτησή σας. Έχει να κάνει με την ποικιλία της Ευρώπης και με την ποικιλομορφία των στόχων, ομάδων στόχων, ενώ η προηγούμενη ερώτηση επιτρέψτε μέσα το επαναλαμβάνω για να είναι πιο καθαρά για μα και για τις ομιλήτρε. Η προηγούμενη ερώτηση τη βοηθού του κ. Ταραμπέλα έχει να κάνει με τις δυνατότητες, τις περιορισμένες δυνατότητες που έχει ένας βουλευτής να κάνει τα μέσα ενημέρωσης, κυρίως τα γυναικεία περιοδικά, να ενδιαφερθούν για το έργο μα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τρίτη ερώτηση. Υπάρχει. Τρίτη ερώτηση. Σχολιασμός. Μπαλντούτσι, μια ερώτηση σχετικά με κάποιες τεχνικές στις οποίες αναφερθήκατε στις παρουσιάσεις σας. Δηλαδή η χρησιμοποίηση του χιούμορ και την καταπολέμηση των στερεοτύπων. Και το ερωτώ αυτό από πλευράς των γυναικείων υποψηφίων στις εκλογές οι οποίες παρουσιάζονται στις εκλογές. Υπάρχει κανένα μειονέκτημα για τις γυναίκες να σου πείσουν αυτά τα, αυτές τις τεχνικές υπάρχει κάποιος κίνδυνος, αν έχουν κάποιο κίνδυνο. Σκέφτομαι τις γερμανικές ε, εθνικές εκλογές. Ε, Άγγελα Μέρκελ και άλλοι ηγέτες ε, προσπάθησαν να χρησιμοποιήσουν το χιούμορ και πρόθεσαν κάποια πράγματα μέσω του ίντερνετ τα οποία ναι μεν έτυχαν της προσοχής των ε, μέσων ενημέρωσης αλλά δεν αποτέλεσαν ένα ικανοποιητικό μέσο για την πολιτική του εκστρατεία. Ρωτώ λοιπόν υπάρχει κάποιος κίνδυνος ενδεχομένω να χρησιμοποιήσει κανείς χιούμορ και να αγωνιστεί κατά των στερεοτύπων σε αυτές τις περιπτώσεις. Πολύ. Άλλη παρέμβαση από κάποιον άνδρα ίσως. Έχει σημασία να δούμε πώς τα ερεθίσματα που πήραμε οι γυναίκες και οι άνδρες από αυτές τις παρουσιάσεις. Όχι, δεν βλέπω να υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον. Οπότε έχουν το λόγο οι ομιλήτρες να απαντήσουν, να συμπληρώσουν για να αξιοποιήσουμε όσο δυνατόν περισσότερο ε, το ενδιαφέρον και το πνεύμα, όχι μόνο τις συγκεκριμένες απορίες, αλλά και το πνεύμα που έχετε καταλάβει ότι υπάρχει διάχυτο στην αίθουσα. Ε, θα αρχίσει η κυρία Ντεβός ή η κυρία Να απαντήσω στο πρώτο ερώτημά σας. Πώς μπορούμε να προκαλέσουμε το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωση. Η απάντηση βρίσκεται στην παρουσίασή μου. Ήταν ο δεύτερος κανόνας να φροντίσουμε να είμαστε συνεπείς. Αν θέλετε να ανακοινώσετε τον ρόλο που παίζετε στην κοινωνία, θα πρέπει να το, προ... να το προβάλλετε με τέτοιο τρόπο ώστε τα μέσα ενημέρωσης να ενδιαφερθούν. Προσπαθούν να ενημερώσουν το κοινό σχετικά με τα τεκτενόμενα και αν η ιστορία σας είναι σημαντική και στοχευμένη, τότε είμαι σίγουρη πως τα μέσα ενημέρωσης θα γράψουν το ζήτημα και θα το παρουσιάσουν. Και κάτι ακόμα. Εάν ε, επικοινωνείτε, πρέπει να επικοινωνείτε ως άτομο, ως πρόσωπο, όχι ως θεσμός. Διαφορετικά δεν ε, πρόκειται να ε, αποκτήσετε την προσοχή των μέσων και των πολιτών. Τώρα, οι πολιτικές διαφορές. Σας ε, ανέφερα τρία, τρεις περιπτώσεις ε, κοινωνιών ε, σε ό,τι αφορά το θέμα χάρη της διαφοράς των αμοιβών. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχουν κάποιες εκστρατείες όπως οι οι αμοιβές που μπορούν να λειτουργήσουν παντού. Τώρα, το θέμα εκεί που σας έδειξα για, με τις προσβολές εντός της εταιρείας κλπ. Αυτό όμως ε, δείχνει ότι υπάρχει μια νέα τάση η οποία μας επιτρέπει να έχουμε μια πολύ καλύτερη επαφή και επικοινωνία. Πρέπει να μπορέσετε να γίνετε κατανοητοί, οι κατανοητές, να στέλνετε μεν γενικά μηνύματα, αλλά να προσπαθήσετε για κάθε χώρα να ε, δουλέψετε πάνω στο facebook, ή στα διάφορα blog, όλα αυτά φυσικά εξαρτώνται και από τα μέσα που χρησιμοποιήσετε. Αλλά υπάρχουν κάποια γενικά στοιχεία που μπορείτε να χρησιμοποιείτε. Και τρίτη ερώτηση, εάν και κατά πόσο κινδυνεύουμε χρησιμοποιώντας χιούμορ. Ε, αυτό νομίζω βρίσκεται στο DNA σας το χιούμορ. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σύμφωνα με το DNA σας. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Εάν όμως δεν σας βγαίνει, παρακαλώ μην το κάνετε. Πρέπει λοιπόν να είστε ειλικρινείς και συνεπείς με τον ίδιο σας τον εαυτό. Να είστε λοιπόν έντιμοι με τον εαυτό σας και όταν επικοινωνείτε να βάζετε τον εαυτό σας, να βάζετε όλη σας ε, την πυθό ακόμα και αν δεν έχετε χιούμορ, μπορείτε να πείτε ένα ανέκδοτο, να πείτε ένα αστείο. Εντάξει, εγώ δεν έχω χιούμορ, λέω ένα ανέκδοτο, πολλές φορές ε, περνάει. Επαναλαμβάνω λοιπόν τώρα τον εαυτό μου, όταν επικοινωνείτε να είστε ο ίδιος ο εαυτός Μην υποκρίνεστε με λίγα λόγια. Ευχαριστώ πολύ. de Paul de ce matin qui a cassé le... Κάποιος ε, χάλεσε το μικρόφωνο σήμερα το πρωί. Λοιπόν, να απαντήσω στις ερωτήσεις τώρα. Στο ζήτημα το, να προκαλέσουμε το ενδιαφέρον και των μέσων ενημέρωσης θα πρέπει φυσικά να μπορείτε να κατανοείτε το κοινό και να στοχεύετε το κατάλληλο μέσο ανάλογα με τα θέματα που θέλετε να προωθήσετε. Λοιπόν, σε μερικές περιπτώσεις ε, αυτό το οποίο κάναμε είναι ήρθαμε σε εποφή με εκδότες γυναικείων περιοδικών για να δούμε πώς ε, θα μπορούμε να προωθήσουμε κάποια χαρακτηριστικά κλπ. Και αν θέλετε λοιπόν να προωθήσετε το θέμα σας σε ευρύτερο κοινό, αυτό αναφίβολα θα μπορούσε να γίνει μέσω των, του εξοικευμένου αυτού τύπου. Επίσης μπορούμε να... Καλέσαμε μάλλον γυναίκες δημοσιογράφους σε δύο περιπτώσεις. Τους δώσαμε λοιπόν κάποια παραδείγματα, δώσαμε και ενδεχόμενα κάποια δείγματα προϊόντων κλπ. Και, και τους είπαμε κοιτάξτε δοκιμάστε το αυτό και θα δείτε την αποτελεσματικότητά του. Φυσικά ήταν ε, ε, πολλές οι οποίες ε, επιθυμούσαν να κατανοήσουν περισσότερα πράγματα π.χ. πώς λειτουργεί η μόδα και άλλα. Το ζήτημα είναι να μπορείτε να στοχεύετε τους ε, κατάλληλους δημοσιογράφους ε, με τον κατάλληλο τρόπο. Τώρα, οι διαφορές. Ε, αυτό είναι κάτι που επανέρχεται ειδικά στο πλαίσιο των μεγάλων διαφημιστικών εκστρατιών. Υπήρξε μια πολύ μεγάλη τάση για τη διεθνοποίηση αυτών των εκστρατιών και πολλές έρευνες έγιναν σχετικά με τις πολιστικές διαφορές και κατά πόσο μπορεί να εφαρμόσετε μία εκστρατεία που να ισχύει σε διάφορες αγορές. Ε, γενικά μπορείτε, εάν φυσικά μπορέσετε να πάρετε ε, τα θέματα που αφορούν την κοινωνία της ε, ανθρώπινες αλήθειες κλπ. Φυσικά υπάρχουν διαφορετικές ευαισθησίες π.χ. υπάρχουν κάποια πράγματα αυτά που σας έδειξα τα οποία δεν ε, έδειξα στι χώρες της Μέσης Τώρα, για το χιούμορ. Ε, θυμάμαι τον Τόνι Μπλερ όπου κάπου τον είχαν δείξει πως ήταν έγκυος τότε πραγματικά ήταν ε, τεράστιο τεράστια το αντίκτυπο ένα άνδρας έγκυο. Έχουν περάσει εδώ και 15 χρόνια από τότε. Αλλά διερωτώ με κατά πόσον αν ε, κανεί ε, διακινδυνεύει ε, χρησιμοποιώντα το χιούμορ. Ναι, εντάξει, αν δεν σα βγαίνει, όπω ακούστηκε και πριν, μην το χρησιμοποιήσετε το χιούμορ. Αν δεν έχετε χιούμορ και φλέγμα, μην το χρησιμοποιείτε. Αναφέρατε την περίπτωση της Άγγελα Μέρκελ. Υπάρχει κάποια αντίδραση από το ακροατήριο. Όχι. Λοιπόν, εδώ τελειώνει και αυτή η ενότητα, αλλά τελειώνει και η μερίδα που μας έχει φέρει όλους μαζί σήμερα. Ε, τελείωσε, πιστεύω, πολύ δημιουργικά, διότι ε, ακούστηκαν πράγματα τα οποία ε, μπορούν να αποτελέσουν μια πλατφόρμα για να χρησιμοποιήσουμε ε, αυτά τα οποία παράγουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να τα χρησιμοποιήσουμε σαν εργαλεία, ε, όχι μόνο προβολής του δικού μας έργου, γιατί ο κάθε βουλευτής έχει και αυτό το, την πρόκληση να προβάλλει τη δική του δέσμευση, τη δική του παραγωγή έργου, αλλά να τα χρησιμοποιήσουμε και σαν εργαλεία για να φέρουμε την Ευρώπη πιο κοντά στις γυναίκες και τις γυναίκες πιο κοντά στην Ευρώπη. Είναι αλήθεια ότι ο τομέας αυτός έχει πολλές ιδιαιτερότητες, διότι είδαμε ότι οι γυναίκες διακατέχονται από κάποια ειδικά αισθήματα, ειδικέ απόψεις ε, για τη θέση τους στην κοινωνία, για την ε, ε, ασφάλεια, την προσωπική τους. Ήδη μας δώσατε παραδείγματα που δείχνουν ότι χρειάζεται μια ειδική προσέγγιση. Χρειάζονται μια ειδική προσέγγιση γυναίκες. Εγώ θα έλεγα ότι αν ασχολούμεθα ιδιαίτερα και με το πώς θα πλησιάσουμε τους άνδρες θα ανακαλύπταμε και εκεί οι ιδιαιτερότητες. Αλλά ας μείνουμε σε αυτές τις ιδιαιτερότητες των γυναικών. Είναι λοιπόν μια αφορμή η σημερινή μας συζήτηση που δεν μπορεί να καλύψει όλες τις παραμέτρους διότι βλέπουμε ότι χρειάζεται και, χρειάζονται και εργαλεία επικοινωνίας, χρειάζονται και γνώσεις ψυχολογίας, χρειάζονται και γνώσεις ε, επικοινωνίας τόσο του βουλευτή τόσο των θεσμικών μας οργάνων, όσο και του, και του staff του βουλευτή. Ήταν πολύ ενδιαφέρον ότι είχαμε την παρέμβαση της βοηθού βουλευτή που ασχολείται με την, ε, με την πρόθεση της ε, πολιτικής υπέρ των γυναικών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ένα σύνολο λοιπόν παραγόντων, ένα σύνολο προκλήσεων, αλλά πιστεύω ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε και εμείς α, ε, α, ως βουλευτές ε, και οι εκπρόσωποι του, του οργάνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι εκπρόσωποι της ε, Γενικής Διεύθυνσης Πληροφόρησης, ότι αξίζει τον κόπο να ασχοληθούμε ιδιαίτερα, διότι όσο περισσότερο προβάλλουμε αυτά που κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τις γυναίκες, τόσο περισσότερο φέρνουμε τις γυναίκες πιο κοντά ε, στην Ευρώπη, τόσο περισσότερο δηλαδή κάνουμε την κοινωνία και την πολιτική συμμετοχική και τόσο περισσότερο τα αποτελέσματα θα είναι αυτά που θέλουμε. Να αισθάνονται πολίτες της Ευρώπης και οι άνδρες και οι γυναίκες. Και στην πλευρά των γυναικών νομίζω ότι έχουμε να δουλέψουμε ακόμη περισσότερο. δύναμή μας είναι η πίστη μας ότι οι γυναίκες αποτελούν ένα σπουδαίο ανθρώπινο δυναμικό σε αυτή την προσπάθεια για μια Ευρώπη αποτελεσματική, ειρηνική, παραγωγική και από την άλλη πλευρά ότι αυτά που έχουμε πετύχει σε συνεργασία ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο είναι ήδη ορατά και αρκετά. Μένει να τα αξιοποιήσουμε μαζί μετά με τις μεθόδους που σήμερα ήδη αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε ότι θα είναι χρήσιμες στο έργο μας, αρκεί λοιπόν να αξιοποιήσουμε τα επιτεύγματά μας για να πείσουμε την ευρωπαϊκή κοινωνία ότι η Ευρώπη είναι μια προστιθεμένη αξία στη ζωή τους και να φέρουμε και τους πολίτες πιο κοντά στο έργο μας. Όσο περισσότερο μας παρακολουθούν, τόσο περισσότερο αντιλαμβάνονται αυτό που κάνουμε, τόσο περισσότερο η διάδραση γίνεται πιο ζωντανή και αμφίδρομη. Και θέλω να ευχαριστήσω θερμά τη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας και Πληροφόρησης για τη σημερινή εναρκτήρια εκδήλωση, ιδιαίτερα τη Διευθύντρια την κυρία Ομπερχάουζερ, τον κύριο Νανσί, που είχαν και την καλή διάθεση να μείνουν μέχρι τέλους μαζί μας και πιστεύω ότι η στιγμή αυτή, η φετινή παγκόσμια ημέρα της ε, γυναίκας, έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ένας πιο δυνατός πολιτικός παράγοντας.